Uh, Ας ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι την ε, συνεδρίασή μας, την κοινή αυτή κοινοβουλευτική συνεδρίαση που θα ασχοληθεί με το σημαντικότατο ενεργειακό ζήτημα και θα αρχίσω να μιλώ στη μητρική μου γλώσσα, την πολωνική και θα μπορείτε να ακούτε τη διερμηνία σε 21 γλώσσες 22η είναι η μητρική μου. Θα υπάρχει διερμηνία και προς πολωνικά. Δεν έχουμε μαλτέζικα σήμερα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε λοιπόν τα ακουστικά σας και σας δίνω χρόνο να τα πάρετε, να τα φορέσετε για να μπορέσω να αλλάξω και να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να καλωσορίσω μάλλον τον κύριο Φρανθίσκο Χαριέρ Ρόχο Γκαρθία, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα και ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Γερουσίας, του, ή μάλλον της Γερουσίας της Ισπανίας και συνδιοργανώνεται αυτή η συνεδρίαση συνδιοργανωνεται αυτη η συνεδρία απο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ισπανική Προεδρία. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από τις υποψήφιες χώρας. Έχουμε και δύο βασικούς ομιλητές. Θα πάρουν το λόγο. Την κυρία Λί Χάντσα, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Τίλμπερκ και ο κύριος Μάρκ Φαντερβάλτερ, που είναι καθηγητής του δικαίου ανταγωνισμού στο Πανεπιστήμιο Έρασμος του Ρότερνταμ και είναι καθηγητής και στο King's College του Λονδίνου. Έχουμε και εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, τον κύριο Πέντρο Λουίς Μαρίν Ορίμπε, υπουργό στο Υπουργείο Εμπορίου και Ενέργειας, υφυπουργό του Υπουργείου Ενέργειας και Εμπορίου της Ισπανίας, Καλωσορίζουμε όλες τις ανταλλαγές απόψεων με το Συμβούλιο, την Προεδρία και, έχουμε και τον κύριο Γιωακή Μαλμούνια που είναι Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας καλωσορίζουμε θερμά και σας κύριε Επιτροπέ. Θα συμμετάσχουν όλοι αυτοί που σας παρουσίασα στη συζήτηση που θα γίνει αύριο. Θα έχουμε και πολλούς συμβούλους και βοηθούς που είναι παρόντες, έχουμε και επισκέπτες ε, πάνω στα θεωρία του κοινού. Χαιρόμαστε πάντα να βλέπουμε παρατηρητές που παρακολουθούν τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι λίγο πιο ψηλά από εμά στα θεωρία που ότι είμαστε εμείς εδώ στην αίθουσα. Ευχαριστώ που ήρθατε για να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι μία από τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας είναι η κοινή ενεργειακή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που είναι εξαιρετική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η συνεδρίαση εκφράζει το πόσο σημασία δίνουμε σε αυτή την προτεραιότητα της Ισπανικής Προεδρίας. Κατά τη διάρκεια σημερινής ε, συνεδριάσεως θα προεδρεύω μαζί με τον πρόεδρο του Ισπανικού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω, τον πρόεδρο του Ισπανικού Κοινοβουλίου, για το πνεύμα συνεργασίας που επεκράτησε την προετοιμασία της συνεδριάσεως. Οι διακοινοβουλευτικές αυτές συνεδριάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι μπορούν να συμμετέχουν στα κοινοβούλια. Κάτι που ήταν και πρόθεση άλλωστε της συνθήκης της ε, Λισαβόνας θα διαρκέσει δύο ημέρες η συνεδρίασή μας, σήμερα και αύριο και έχετε λάβει όλοι σας πρόγραμμα της διακοινοβουλευτικής αυτής συνεδριάσεως με θέμα της μελλοντική ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πώς θα διαμορφωθεί και πώς θα δώσουμε δυνατότητες ανάπτυξη επιχείρησής μας. Πώς η διαδικασία αποφάσεως, αποφάσεων των κρατών μελών θα διαπνέεται από μια συνέπεια θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι οι πολίτες μας θα αισθάνονται τις θετικές συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνουμε. Ο κόσμος έχει προσδοκίες όσον αφορά τον εφοδιασμό σε ενέργεια, έχει μεγάλες προσδοκίες και θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Θα δώσω το λόγο τώρα στον πρόεδρο της Γερουσίας της Ισπανίας, τον κύριο Φρανσίσκο Χαβιέρ Ρόχο Γκαρθία. Και ίσως κύριε Πρόεδρε θα μπορούσατε να κάνετε κάποια εισαγωγικά σχόλια. Έχει το λόγο. Καλό σας απόγευμα. Εξοχότατε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι συνάδελφοι Ευρωβουλευτές και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα να έχω την ευκαιρία να σας προσφωνήσω στην ολομέλεια αυτού του θεσμικού οργάνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερίδων που θα είναι συνάντηση μεταξύ των ε, εθνικών βουλευτών και των ευρωβουλευτών για να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε για ένα θέμα που είναι τόσο επίκαιρο και τόσο σημαντικό όπως η ενεργειακή πολιτική του 21ου αιώνα. Η συνάντηση που ξεκινάει τώρα είναι μια απόδειξη ακόμα παραπάνω για την αναγκαία συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων προωθώντας ε, τους μηχανισμούς ε, μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας προς αυτό το στόχο. Η ενεργειακή πολιτική που επικεντρώνουμε τη συζήτησή μας αυτή σήμερα είναι μια πολιτική που και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ικανότητα που θα καταδείξουμε για να ανανεώσουμε τις παραγωγικές μας δομές και να κάνουμε για την Ευρώπη και κάθε μια από τις χώρες που τη συναπαρτίζουν ανταγωνιστικές οικονομίες με αηφορία στην δράση τους. Αυτή η τοποθέτηση που πριν από κάποια χρόνια μπορούσε να θεωρηθεί ένας επενέσιμος στόχος, σήμερα έγινε ανάγκη πλέον, αναγκαιότητα. Και αν το επιτρέπετε, κιόλα πιέζει ο χρόνος και είναι κατεπήγον το θέμα υπό τους οικονομικούς όρους ε, για τη ε, διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε και στη συγκυρία που βρισκόμαστε υποχρεώνεται η Ευρώπη και κάθε μια από τις χώρες της να συνεργαστούν όλοι ώστε να δημιουργηθεί ο χώρος ε, που θα είναι η καλύτερη εγγύηση για την ευημερία που μπορούμε να αφήσουμε στις μελλοντικέ γενναίες. Σε αυτή την τάξη των πραγμάτων η ενεργειακή πολιτική είναι μια σημαντική συνιστόσα επί της οποίας πρέπει να στηριχθούμε και να οικοδομήσουμε τις πολιτικές για το μέλλον. Και αφενός ε, βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε οι ευρωπαϊκές οικονομίες να ξεπεράσουν το δυνατόν ταχύτερα την κατάσταση που στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή που είναι μια κατάσταση ε, στασιμότητας και πρέπει ταυτόχρονα να δημιουργηθούν οι βάσεις ε, για να αποκτήσει η ευρωπαϊκή οικονομία τα αναγκαία μέσα για να έχει ένα υφόρο πρότυπο, ισορροπημένο, ισόρροπο πρότυπο και ανταγωνιστικό. Ω προ αυτόν τον στόχο είναι θεμελιώδε τα θεσμικά όργανα και οι κυβερνήσει Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστούν από κοινού για να αρθρώσουν προγράμματα και σχέδια και μέτρα που στον ενεργειακό τομέα θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα, την ε, ασφάλεια στην ε, κάλυψη των αναγκών λαμβάνοντας υπόψη βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. στόχους. Πρώτα απ' όλα αυτή η σημαντική προσπάθεια πρέπει να επικεντρώνεται ώστε βήμα προς βήμα σταδιακά να υπάρξει διασύνδεση ενεργειακή μεταξύ των κρατών μελών ώστε να υπάρξει ένα σταθερό δίκτυο ενέργειας στην Ευρώπη που θα προωθήσει την ενιαία εσωτερική αγορά. Ένα σταθερό μόνιμο δίκτυο που θα πρέπει να ολοκληρώνεται και να συμπληρώνεται με τα συστήματα και σχέδια διασύνδεση με τα ε, όμορα κράτη, με τα γειτονικά κράτη. Επίσης πρέπει να προχωρήσουμε στην αποδοτικότητα ενέργειας ε, στις επιδόσεις μας, κάνοντας χρήση καθαρών πηγών ενέργειας, ώστε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από εισαγόμενους πόρους ε, ενεργειακούς, βελτιώνοντας την πολιτική μας και έτσι βαθύνοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Στο παρελθόν είχαμε τριβές και η σπανίδα των ενεργειακών πόρων είχε οδηγήσει σε τριβές και προβλήματα μεταξύ κατών μελών. Τώρα θα πρέπει αυτή η τάση να πάψει να ισχύει. Η ε, νέα ύπαρξη νέων πηγών καθαρών και ανεξάντλητων ανοίγει μια νέα προοπτική ευημερία και ειρήνης. Γι' αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να υπάρξουν κοινοτικέ διατάξει και ρυθμίσει ω προ αυτά τα θέματα, δράτω με τι ευκαιρίε τη παρουσία των ε, μελών των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων ώστε να εμβαθύνουμε σε αυτέ τι πτυχέ και να εκπονήσουμε δημιουργήσουμε προγράμματα εθνικά τα οποία θα συγκλίνουν με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να προαχθούμε προς την κοινή ίδια κατάσταση, ε, κατεύθυνση. Αυτό το χρειάζεται η Ευρώπη και εμεί το χρειαζόμαστε ώστε στη γυραιά ήπειρο της Ευρώπης να δώσουμε τη δυνατότητα να ευδοκιμήσουν οι ελπίδες τον 21ο ε, αιώνα και οι προσδοκίε των Ευρωπαίων. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ευρωβουλευτέ, ε, γι' αυτό ευθύνη μας είναι από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το Εθνικό Κοινοβούλιο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ να εργαστούμε ώστε να υπάρξει η Ευρωπαϊκή Ενιαία Εσωτερική Αγορά για τα ενεργειακά θέματα που θα είναι ασφαλής, θα είναι μόνιμη και θα σέβεται το περιβάλλον. Θα βοηθήσει τους βιομηχανικούς τομείς μας και τους πολίτες μας ώστε να διασφαλίσουν την ευημερία και την κοινωνική συνοχή. Έτσι ελπίζω και αυτό προσδοκώ ότι θα γίνει. Και αυτές οι ημερίδες θα είναι επίκεντρο αυτών των συναντήσεων και του προβληματισμού ώστε όσα θα εξετάσουμε να προσεγγίσουμε στο εγγύς μέλλον να γίνουν πραγματικότητα. Διότι αυτή η πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο θα αφήσουμε ω κληροδότημα στις μελλοντικέ γενναίες. Και εκείνοι θα μπορέσουν καλύτερα από εμά να υλοποιήσουν και να δρέψουν τους καρπούς από αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό εγχείρημα το οποίο οικοδομούμε, που είναι η μεγαλύτερη μεγάλη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτή την εισαγωγική σας παρέμβαση. Ευχαριστώ και πάλι. Ε, κυρίες και κύριοι, πριν προχωρήσουμε και πάμε στην παρουσίαση των εμπειρογνωμόνων μας, θα ήθελα να πω ένα-δύο πράγματα εν είδη εισαγωγή στη συζήτησή μας. Και αυτό θα βασιστεί στα όσα μας είπε ο πρόεδρος της Γερουσίας της Ισπανίας. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μεγάλη πρόκληση όσον αφορά την ολοκλήρωση της ε, κοινή αγοράς, της ενιαίας αγοράς. Η ενιαία αγορά είναι ένας τρόπος να ε, αναπτυχθούμε και να βγούμε από την κρίση. Αναφέρομαι βέβαια στην οδηγία περί υπηρεσιών. Αναφέρομαι στην ε, τυποποίηση, την έλλειψη μάλλον της τυποποίησης, που σημαίνει ότι δεν έχουμε πραγματικά ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων. Θα πρέπει και οι καρποί της έρευνας να κινούνται ελεύθερα, μαζί βέβαια με, τα, με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Άλλο ένα θέμα είναι η κοινή ενεργειακή αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι μια ισχυρή ενεργειακή κοινότητα στο μέλλον. Αρκεί μόνο να συγκρίνει κανείς τη δική μας κατάσταση με αυτή της Κίνας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι για να πετύχουμε εμείς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων μας θα πρέπει να κινηθούμε ως κοινότητα στην παγκόσμια αγορά. Έτσι, πριν από δύο εβδομάδες περίπου, με τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ζακ Ντελόρ, που ήταν πρόεδρος από το 1984 μέχρι το 1994, ζητήσαμε να δημιουργηθεί μια νέα κοινότητα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας. Αυτό θα θέλαμε να πραγματοποιηθεί εντός των ισχυουσών δομών των συνθήκων. Ε, δεν θέλουμε κάτι που θα είναι εκτός της δομής της συνθήκης, χωρίς να το αποκλείουμε αυτό. Όμως, για πρώτη φορά η συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρεται σε ενεργειακή αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αναφέρεται και σε κοινή πολιτική στον τομέα. Είναι μια νέα ιδιότητα, νέα ποιότητα, ένα νέο χαρακτηριστικό της συνθήκης της Ένωσης και θα πρέπει να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτό το νέο χαρακτηριστικό. Οι λαοί της Ευρώπης θέλουν ε, ενέργεια που να είναι σε λογικές τιμές είναι θέμα οικονομίας κλίμακας. Έχουμε μια μεγάλη σημαντική ευρωπαϊκή αγορά και αν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε την αγορά αυτή σαν ένα σύνολο, τότε θα είναι φθηνότερη ενέργεια. Φθηνότερος εφοδιασμός ενέργεια. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αφορούν την αλλαγή του κλίματος. Μέχρι 80% των, της αλλαγής του κλίματος οφείλονται ε, στην ενεργειακή, στη χρήση της ενέργειας. Μόνο 20% της αλλαγής του κλίματος οφείλεται στη χαλιβουργία, στη χημική βιομηχανία, ε, στην παραγωγή τσιμέντου κλπ. 80% των προβλημάτων στον τομέα του κλίματος 80% ε, των προβλημάτων μπορούν να επιληθούν μέσω ενεργειακής αντιμετωπίσεως. Πρέπει να υποστηρίξουμε επίσης τους τις μεγάλες επιχειρήσεις ενέργειας, τους γίγαντες. Θα πρέπει να μπορούν να επενδύσουν σε μακροχρόνια βεβαιότητα στον εφοδιασμό ενέργειας. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας βέβαια και θα πρέπει να ανταποκριθούμε και στις ε, προσδοκίες των πολιτών μας. Μία ενεργειακή κοινότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη αποφασίσαν να υπογράψουν μια χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλα τα συμβαλόμενα μέρη, τα συμβαλόμενα κράτη θα δεσμευτούν να ακολουθούν μια κοινή πολιτική. Και να προωθούν σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, εφαρμόζοντας και ισχύουσα νομοθεσία. Διότι δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά όλες οι ισχύουσες ε, νομοθεσίες όπως το δεύτερο και τρίτο ενεργειακό πακέτο. Το δεύτερο ενεργειακό πακέτο υιοθετήθηκε από την Ένωση πριν από μερικά χρόνια. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτές τις αποφάσεις. Οπότε θέλουμε αποτελεσματική υποστήριξη των πολιτικών και κάποια συγκεκριμένα βήματα αν αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Οι εμπειρογνώμονές μας θα αναφερθούν σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν διάφορες επιλογές όσον αφορά τις που προσφέρει ο Ευρωπαϊκός Νόμος και οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν κλείνω καμία πόρτα. Το μόνο που λέω είναι ότι ακόμα και χωρίς αλλαγή των συνθήκων υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και εν κατακλείδη έχω τέσσερις προτάσεις να κάνω. Τέσσερις τομείς να αναφέρω που νομίζω θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε στον τομέα της ενεργειακής ε, πολιτικής Πρώτα απ' όλα θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε τα βιομηχανικά μας δίκτυα, τις δυνατότητες αποθήκευσης και να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα δίκτυα αποτελεσματικά ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ασφαλή εφοδιασμού ε, ασφάλεια εφοδιασμού ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου κλπ. σε περίπτωση ανάγκης, όλες τις μορφές ενέργειας. Η οδηγία για το φυσικό αέριο Υποτίθεται ότι κάνει ακριβώ αυτό. Είναι επιτάπητο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υποτίθεται ότι θα μα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε κρίσει. Δεύτερο τομέα κοινή έρευνα, η έρευνα, έρευνα σε μεγάλη κλίμακα. Διότι χρειαζόμαστε νέε τεχνολογίε, νέε λύσει σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, εξοικονόμηση ενέργεια, πιο αποτελεσματική παραγωγή και πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας από πλευράς τελικού χρήστη. Και θα πρέπει να τα καταφέρουμε όλα αυτά μειώνοντας ταυτόχρονα τις εκπομπές των ορυκτών καυσίμων, διότι θα χρησιμοποιήσουμε επί πολλά χρόνια ακόμα τα ορυκτά καύσιμα και θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η τεχνολογία ε, σύλληψη, συλλογή άνθρακος και αποθήκευσης άνθρακος είναι κάτι που μπορεί να μας εξυπηρετήσει. Και τρίτος τομέας κοινής δράσης θα μπορούσαμε να συναθρήσουμε τις δυνατότητες αγοράς που έχουμε. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίζει με, μεζί με μεγάλες, μεγάλους βιομηχανικούς φορείς εισαγωγή ενεργειακών πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ώρα διάφορα κράτη-μέλη, διάφορες εταιρείες αγοράζουν ξεχωριστά από τους ίδιους προμηθευτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ανταγωνιζόμαστε ένα τον άλλον. Και αυτό οδηγεί σε εντάσεις μεταξύ των κρατών μελών και σε αποδυνάμωση μιας κοινή ε, ισχύω τα λέγαμε, του δυνατού μας σημείου. Ναμπούκο, South Stream, North Stream, Yamal, ε, Amber. Έχουμε πάρα πολλές συζητήσεις που διεξάγονται όσον αφορά αυτά τα θέματα, αλλά θα πρέπει να μειώσουμε τις εντάσεις που υφίστανται. Και τέταρτος τομέας δράσης πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε, το πώς χρησιμοποιούμε την ενέργεια. Ο τρόπος ζωής μας θα πρέπει να αλλάξει. Χρειαζόμαστε πραγματικά να εξοικονομήσουμε ενέργεια και αυτό είναι δουλειά των κρατών μελών, των κυβερνήσεων, είναι δουλειά των εθνικών κοινοβουλίων. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να κλείσω τονίζοντας ότι μόνο Εάν τα εθνικά κοινοβούλια και εθνικέ κυβερνήσει ενδιαφερθούν για μια κοινή πολιτική, μόνο συμφωνούμε όλοι ότι είναι κάτι που αξίζει τον κόπο και αν συμφωνήσουμε όλοι ότι αξίζει τον κόπο για τους πολίτες μας, τότε η ενεργειακή κοινότητα θα μπορούσε να δει το φως της ημέρας, θα μπορούσε να λάβει διάφορες μορφές, υπάρχουν διάφοροι δρόμοι που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Αλλά μόνο αν κινηθούμε όλοι μαζί θα μπορέσουμε τελικά να νικήσουμε τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι δουλειά μας τώρα να σχεδιάσουμε, να σχεδιάσουμε αυτή τη μελλοντική κοινότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ και να δώσω το λόγο στους φιλοξενούμενους μας ομιλητές. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον κύριο Μάρκ Φαντερβάλτερ, καθηγητή ενεργειακού δικαίου στο King's College του Λονδίνου και τον καθηγητή ανταγωνισμού στο Πανεπιστήμιο Έρασμος του Ρότερνταμ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του συναδέλφου Λί Χένσερ που κάθεται εδώ, ε, θα πρέπει να σας πω ότι είναι τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ και να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη μας για την ενεργειακή κοινότητα, αν θέλετε. Σας έχουμε δώσει κάποιες διαφάνειες, θα βρείτε τα έγγραφα αυτά τα βασικά στοιχεία της παρουσίασής μας και θα σας ε, παρουσιάσουμε τις διαφάνειες αυτές μία προς μία. Καταρχήν, γιατί κάναμε μία μελέτη για την ενεργειακή πολιτική. Πολλές μελέτες γίνονται τη σήμερα ημέρα. Γιατί, όπως είπα ναι, και οι δύο πρόεδροι, βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, σε μια κρίσιμη φάση όπου θα αντιμετωπίσουμε πιθανότατα μια νέα βιομηχανική επανάσταση και αυτή πιθανότατα θα γίνει στον ενεργειακό τομέα. Αυτό είναι το θετικό στοιχείο αλλά υπάρχουν και κάποια πιο κρίσιμα στοιχεία, όπως η κρίση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, οικονομική, περιβαλλοντική και η εξάρτηση από τις ε, εξωτερικές προμήθειες. Όπως ήδη υπόθηκε λοιπόν, χρειάζεται να κάνουμε κάτι για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Εμείς εξετάζουμε δύο θέματα καταρχήν στην έκθεση. Α, κατά πόσο η Ευρώπη θα είναι στη ηγετική θέση σε αυτή την ενεργειακή επανάσταση ή θα είμαστε ουρακοί και θα ακολουθήσουμε αυτά που κάνουν άλλοι στον υπόλοιπο κόσμο. Και δεύτερη ερώτηση είναι βέβαια ότι το σημερινό σχήμα ενέργειας δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει να ε, κινηθούμε προς μια κοινωνία άνευ άνθρακα. Όπω είπε και ο κύριο Ρόχο Καστίγια, χρειάζεται να ενεργήσουμε επιγόντω. Έχουμε το πρόγραμμα 2020 για, 10, για τα επόμενα 10 χρόνια. Άλλε χώρε ήδη κινούνται, η Κίνα, η ΕΠΑ, πιο γρήγορα από εμά. Θέλουμε να του προλάβουμε και υπάρχει και μια πιεστική ζήτηση από την βιομηχανία. Ήδη κινείται η βιομηχανία και χρειάζεται να ενεργήσουν και οι πολιτικοί. Η μελέτη μα, ωστόσο, δεν αφορά την πολιτική. Είναι απλά νομική, αφορά το νομικό πλαίσιο και προσφέρει τι επιλογέ που η πολιτική πολιτική, εσείς δηλαδή, είτε είστε στα Εθνικά Κοινοβούλια είτε στο Ευρωκοινοβούλιο, πολιτικές που εσείς μπορείτε να αποφασίσετε. Έχουμε χειριστεί αυτό το νομικό ζήτημα σε, τρεις υπο, ε, σε τρία υποερωτήματα. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε στην έκθεσή μας είναι γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί ήδη υπάρχει ενεργειακή πολιτική ευρωπαϊκή και έχουμε και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τι δεν πάει καλά λοιπόν με το ισχύον σύστημα. Αν κάτι δεν πάει καλά, τι πρέπει να γίνει, ποια είναι τα μέτρα πολιτικής που μπορούμε να προβλέψουμε και τέλος ποια είναι τα νομικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να επιτύχουμε τα μέσα αυτά που θα χρειαστούμε για να βελτιώσουμε τις πολιτικές μας. Το πρώτο ερώτημα το οποίο θα με το οποίο θα ασχοληθεί ο καθηγητής Χέντζη αφορά το ισχύον νομικό σύστημα. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο εγώ εξέτασα είναι αν υπάρχει ενεργειακή πολιτική, αν υπάρχουν δηλαδή τα νομικά μέσα για να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική και η απάντηση είναι εν μέρη καλή και εν μέρη κακή. Έχουμε μια συνθήκη του Ευρατόμου υπέρ της ενεργείας και ε, ε, η, άλλη συνθήκη που υπήρχε την εποχή της ε, ε, ενώσεως άνθρακα και χάλιβα έχει τώρα εκπνεύσει και τώρα για πρώτη φορά έχουμε εις την γενική συνθήκη τη νέα, ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται ειδικώ στην ενέργεια αλλά το εάν αυτό θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε μια οικονομία με ουδέτερο διεξίδιο του άνθρακος στα πλαίσια τα χρονικά που θέλουμε είναι αμφισβητήσιμο. Εάν κοιτάξουμε λοιπόν τι έγινε τα τελευταία 20-25 χρόνια, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπήρξε μεγάλη ε, ε, δραστηριότητα ε, νομοθετική αλλά ουσιαστικά απέβλεπε στη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτός ήταν ο ουσιαστικός στόχος και μάλιστα ένας στόχος ο οποίος ήταν αυτοσκοπός και όχι ένα μέσον προς ε, την επίτευξη ενός σκοπού. Και μόνο τα τελευταία έτη έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε με άλλους παράγοντες όπως τη δημιουργία την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας για να μειώσουμε την ρήπανση και την κατάρτιση προδιαγραφών για τα κτίρια, για τα πλυντήρια και ούτω καθεξής. Εάν, λοιπόν, αυτά είναι θέματα εσωτερικής αγοράς και αν δούμε πόσο συμμορφώνονται τα κράτη-μέρη τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά διότι έχουμε πάρα πολλές διαδικασίες παραβάσεως στον τομέα αυτό. Το εάν λοιπόν υπάρχει μία ε, ενεργειακή πολιτική αυτή τη στιγμή και αν δούμε πώς οι στόχοι της ισχύουσας πολιτικής έχουν επιτευχθεί βλέπουμε ότι ε, δεν έχουν επιτύχει καλή πρόσβαση στην ισχύουσα πολιτική δεν έχουν ακόμη βιωσιμότητα και από πλευράς πολιτικής ακόμη δεν αποτελούν άρρηκτο μέρος της ΕΝΕΛΚΕ πρέπει ακόμη να ε, ενταχθούν περισσότερο και όσον αφορά την ασφάλεια ε, όπως ήδη ανεφέρθη θα υπάρξει ε, μία νέα οδηγία ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα μέτρα σε περίπτωση κρίσεως. Επαρκεί όμως. Αυτή είναι μία βραχυπρόθεσμη λύση αντίδρασης. Αλλά συνοψίζοντας έχουμε κάνει ορισμένες πρόοδους, όχι όμως επαρκείς. Όπως λοιπόν ελέγχθη, οι τρεις στόχοι έχουν επιμέρους επιτευχθεί, αλλά όχι ε, με συνέπεια και γι' αυτό καταλήγουμε στις ε, τρεις ουσιαστικές ε, απαντήσεις της εκθέσεως ότι δεν υπάρχει συνέπεια, η ενεργειακή πολιτική θεωρείται παράπλευρο θέμα άλλων πολιτικών των κανόνων εσωτερικής αγοράς ή άλλης πολιτικής. Το δεύτερο είναι εάν η πολιτική αυτή μπορεί να αποδώσει γιατί η διαδικασία λήψης αποφάσεως είναι πολύ ε, αργή ενώ χρειαζόμαστε επίγουσα δράση. Δεν υπάρχουν μέσα με τα οποία να κατευθύνουμε την έρευνα και την ανάπτυξη στη σωστή κατεύθυνση ώστε οι επενδύσεις να γίνουν στο σωστό μέρος. Όλοι προσπαθούν να αντιγράψουν τα ίδια πράγματα αλλά χωρίς έναν ουσιαστικό συντονισμό των πολιτικών. Ε, δεν υπάρχει αξιοπιστία. Υπάρχουν πολλές παραβιάσεις από τα κράτη-μέλη και αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που έχουμε διαπιστώσει. Δηλαδή, καταρχήν ε, υπάρχουν αποφάσεις πολιτικές από κυβερνήσεις, από τα κοινοβούλια και μετά παρουσιάζονται στους ενδιαφερόμενους, ενώ θα έπρεπε η διαδικασία να είναι αντίστροφη και οι ενδιαφερόμενοι όπως στις παλιές συνθήκες να εμπλέκονται άμεσα και από την αρχή στην λήψη αποφάσεων. Αν δούμε λοιπόν την παλιά συνθήκη άνθρακος και χάλιβος διαπιστώνουμε ότι έκτοτε υπήρχε μάλλον μία οπισθοχώρηση παρά μία πρόοδο στο θέμα της ενεργειακής πολιτικής. Υπάρχουν πολλοί λόγοι αλλά ορισμένους από αυτούς θα ήθελα να τους αναφέρω. Καταρχήν ότι τα κράτη-μέλη ακόμη θεωρούν ότι η πολιτική τους είναι ε, ε, ε, εθνική και από την άλλη πλευρά η Ευρώπη δεν έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ένα κοινό με το έναντι στους προμηθευτές. Άρα υπάρχει κατακαιρματισμένη πολιτική που δεν είναι συνεπής. Υπάρχει μία συλλογή 27 σχετικά μη αναποτελεσματικών πολιτικών και ε, ζητούμε να είμαστε ε, ε, μέρος στην επόμενη βιομηχανική επανάσταση. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει μία επιλογή. Μία επιλογή να μην κάνουμε τίποτα να μην αναλάβουμε τα φιλόδοξα μέτρα τα οποία χρειάζονται για να προχωρήσουμε οπότε ίσως θα βρεθούμε αντιμέτωποι με άλλη μία κλιματολογική κρίση ή να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπον την κατάσταση, να λάβουμε μέτρα δραστικά. Οπότε, τι τίθεται το ερώτημα, τι δράση και εδώ θα ζητούσαμε εάν ληφθεί ε, δράση να είναι συγκεκριμένη διότι η ενέργεια είναι ζωτική για όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας έχει χαρακτηριστικά που την διακρίνουν από τα άλλα προϊόντα και τις άλλες ε, υπηρεσίες και ε, αυτή τη στιγμή ζητούμε να υπάρχει χαμηλή ανάπτυξη της κατανάλωσης ενεργείας αντί να υπάρχει μία ραγδαία ανάπτυξη. Επίσης οι περισσότερες μορφές ενεργείας πρέπει να μεταφερθούν από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης γι' αυτό και τα δίκτυα είναι πολύ σημαντικά σε αυτό το σημείο. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένες δράσεις όσον αφορά τον τομέα αυτό αυτό αλλά και δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο διότι ε, από πλευράς ευρωπαϊκής ε, ήδη έχουν ε, αναλυφθεί μέσω της συνθήκης Λισαβόνας οι υποχρεώσεις να προχωρήσει το θέμα πιο γρήγορα και δεύτερον υπάρχουν οι ανάγκες που ανέφερε ο πρόεδρος δηλαδή τα κράτη-μέρη θέλουν να προωθήσουν την συνοχή και την αλληλεγγύη και η Ευρώπη πρέπει να μιλά με μία φωνή εις την διεθνή σκηνή δεν πρόκειται για δράσεις μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε, ε, πρόκειται για αποδοτικές δράσεις και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διδαχτούμε από τα λάθη του παρελθόντος να έχουμε ε, ε, <clears throat> πολιτικές οι οποίες να είναι πιο αποτελεσματικές, πιο καλά οργανωμένες, θα επιτρέψουν καλύτερες αποφάσεις και συντονισμό της έρευνας και της ανάπτυξης διότι ε, υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα και τέλος χρειάζεται μια ε, δημοκρατική διαδικασία στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Άρα τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προβούμε σε αποτελεσματικέ επίγουσε ενέργειες. Στην ομάδα εργασία μα εντοπίσαμε δύο είδη μέτρων, καταρχήν τα ουσιαστικά και έπειτα εντοπίσαμε κάποια πολιτική φύση μέτρα, δηλαδή τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να, στα οποία θα πρέπει να προβούν τα θεσμικά όργανα. Όσον αφορά την ουσία, καταρχήν, ακόμα και αν έχουμε εκφράσει επικρίσεις όσον αφορά τις δυνάμεις της αγοράς στην έκθεσή μας, Εν τέλει η Ευρώπη έχει μια ιστορική αγορά, είναι το κεντρικό, ε, ο πυρήνας πάνω στον οποίο ε, βασίζεται η ολοκλήρωση και αναμφίβολα η ελεύθερη αγορά για την ενέργεια θα πρέπει να είναι, ε, παραμείνει ένας από τους βασικούς μας στόχους. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κόμβοι στους οποίους θα συνδέονται όλα τα κράτη-μέλη ώστε να δημιουργείται μια de facto αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη και θα μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σε ένα πιο αποτελεσματικό, με ένα πιο αποτελεσματικό αποδοτικό τρόπο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, η σταθεροποίηση των τιμών ή η εγγύηση των τιμών όταν οι αγορές δεν δίνουν το αποτούμενο αποτέλεσμα αρκετά γρήγορα. Διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ενέργειας της Ένωσης ε, όντα σε θέση να πετύχουμε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ανεξαρτησία ή ασφάλεια ανεφοδιασμού για την Ευρώπη. Αυτό επίσης σημαίνει και αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση επί της ουσίας διαχείριση κρίσεων και κοινό έλεγχο των αποθεμάτων. Και όσον αφορά τώρα τα θεσμικά μέτρα, τους θεσμούς που μπορούν να δώσουν αυτά τα μέτρα και δεν τα αναφέρομαι, αλλά ο κατάλογος των μέτρων δεν είναι ούτως ή άλλως ε, ε, ενδελεχής, μπορούν να προσθεθούν και άλλα μέτρα ε, θα πρέπει να λειτουργήσουν σε συνεργασία με τον βιομηχανία αλλά και τους καταναλωτές γιατί όλοι ενδιαφέρονται για την ενέργεια ε, εκ των προτέρων για, και θα πρέπει να συμμετέχουν στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Να έχουμε έναν ευρωπαϊκό ρυθμιστή, ε, όταν μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό κόμβο ενέργεια που θέλουμε να επιτύχουμε την αλληλεγγύη, θα πρέπει να έχουμε και ένα, μέσο, ε, ένα πυρήνα λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει να μπορέσουμε να, ως Ευρώπη να συντονίσουμε και να ενισχύσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και να έχει την για να σταθεί στη διεθνή σκηνή. Αλλά φυσικά πώς όλα αυτά μεταφράζονται σε νομικό επίπεδο και εδώ μπαίνουμε στην ουσία της έκθεσης. Πρόεδρος διακόπτη. Να αλλάξω τα ονόματά σας εδώ τα καρτελάκια σας γιατί τα έχουμε βάλει ανάποδα. Πρόσεξα. Luckily εμεί ξέρουμε ποιοι είμαστε. Η μεγάλη πρόκληση λοιπόν και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προκλήσεις για τα κοινοβούλια σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την ε, πρόκληση την ενεργειακή θα πρέπει να δούμε τι είδους θεσμικά πλαίσια μπορούμε να σχεδιάσουμε, τι επιλογές υπάρχουν ως προς αυτό και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ίσως με μερικά κράτη-μέλη που μπορεί να θέλουν να προχωρήσουν και πιο γρήγορα από ό,τι άλλα. Ε, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι φυστάμενες δομές της Ένωσης για κάποια που να μπορέσουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Πώς ε, θα ορίσουμε το πεδίο εφαρμογής οποιασδήποτε ενεργειακής πολιτικής, πόσο φιλόδοξη θα πρέπει να είναι αυτή τόσο από την πλευρά της ουσίας όσο και από τη θεσμική άποψη και πώς επιδιώξουμε όλους αυτούς τους στόχους διασφαλίζοντας αυτά που ήδη έχουμε. Το κοινοτικό και εκτιμένο το περίφημο. Την ομολογία, την ομολογία της αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί, τις νομοθεσίες που έχουν αναπτυχθεί εδώ και 60 σχεδόν χρόνια. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Έχουμε λοιπόν τέσσερις βασικές επιλογές για να προχωρήσουμε από θεσμική άποψη. Έχουμε φυσικά την συνθήκη της Λισαβόνας, το 194, το νέο άρθρο που αυξάνει τις αρμοδιότητες της Ένωσης. Επίσης έχουμε την επιλογή της ενισχυμένης συνεργασίας, ε, το άρθρο 20 της συνθήκης, ή να ξεκινήσουμε με μια νέα ενεργειακή συνθήκη. Ε, τέλος, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ρεαλιστική συνεργασία στις ε, γραμμές της συνθήκης ε, του Σέγγεν, ότι δηλαδή επιλέγουμε κάποια σημεία, κάποια θέματα και τα ενσωματώνουμε από αυτής της βάσης. Η πρώτη επιλογή είναι φυσικά η συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, πρόκειται για μια μεγάλη βελτίωση σε σύγκριση με την προηγούμενη ε, συνθήκη όπου η ενέργεια ε, ήταν στην ίδια βάση με τον τουρισμό. Έχουμε δηλαδή μια πραγματική νομική βάση στη συνθήκη. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες αρνητικές πλευρές. Καταρχήν η πρόσβαση στους πόρους και η φορολογία αποκλείονται από τις ε, κανονικές διαδικασίες που ισχύουν σε αυτούς τους τομείς, δηλαδή ε, ισχύει η ομοφωνία για την φορολογία, η αλληλεγγύη δεν ορίζεται ως ένας από τους στόχους και τέλος έχουμε αμφιβολίες όσον αφορά κάποια νομικά εμπόδια που υπήρχαν στις παλαιότερες συνθήκες, όπως για παράδειγμα η, δημιουργία, η δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας, ενός ευρωπαϊκού οργανισμού ενέργειας, ε, η νομολογία μυρώνει, όπως αποκαλείται. Ε, επίσης δεν υπάρχουν εξωτερικές αρμοδιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν οι βελτίωση, αλλά το 194 δεν πιστεύουμε ότι θα δικήσει σε ριζοσπαστικές αλλαγές και ο κατακαιρματισμός θα εξακολουθήσει να ισχύει. Βεβαίως ε, η συνθήκη της Ένωσης έχει αυτή τη δυνατότητα, δίνει τη δυνατότητα για ενισχυμένη συνεργασία όπου εννέα κράτη-μέλη τουλάχιστον μπορούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Αν το θέλουν, αυτή είναι μια βελτίωση που υπήρχε όμως και στην προηγούμενη συνθήκη. Ωστόσο και εδώ οι όροι υπό τους οποίους αυτά τα, νέα, τα εννέα κράτη-μέλη μπορούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα είναι αρκετά βαρύς και φυσικά μπορούμε να εφεύρουμε νέες λύσεις για κάποια νομικά προβλήματα όπως ας πούμε για το ποιος είναι ο ρόλος των θεσμών και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την αυξημένη συνεργασία τα, οι αρμοδιότητες αυξημένης συνεργασίας επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να προχωρήσουν και να κάνουν πλήρη χρήση των θεσμών και στην διεθνή σκηνή. Έχουν επιπλέον νομικές αρμοδιότητες. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Ε, όταν θελήσει κανείς να χρησιμοποιήσει το 194. Είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία. Από νομικής άποψης και όχι από πολιτικής, από νομικής άποψης θα πρέπει να ληφθούν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εντοπίσαμε, να τα βάλουμε σε μια νέα συνθήκη και τη νέα συνθήκη να τη χρησιμοποιήσουμε στη θέση της παλιάς ε, συνθήκης ε, ΕΚΑΧ. Ίσως αυτό να είναι βέβαια όνειρα θερινής νυχτός από πολιτικής άποψης αλλά έχουμε ένα τμήμα της συνθήκης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια παρόμοια ή συγκρίσιμη λύση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μια ε, ε, κοινότητα για την ενέργεια. Θα χρησιμοποιούσαμε δηλαδή το, η βάση της συνθήκης ΕΚΑΧ αλλά για λιγότερα κράτη-μέλη. Είναι ενδιαφέρουσα επιλογή αλλά πιο δύσκολη στην εφαρμογή της. Έχουμε τώρα την πιο ρεαλιστική επιλογή που του να έχουμε έναν οδικό χάρτη για συμφωνίες τύπου Σέγγεν. Και εδώ υπάρχουν διάφορες επιλογές που μπορούμε να εξετάσουμε υπό αυτό το λάβαρο της πιο ρεαλιστικής ε, προσέγγισης. Ας πούμε, ενισχυμένη συνεργασία σε περιφερειακή βάση, να έχουμε διάφορες πλατφόρμες περιφερειακές για να αναπτύξουμε ε, περιφερειακούς κόμβους ενεργειακούς θα μπορούσαμε να έχουμε περιφερειακές συμφωνίες ώστε να συγκεντρωθεί η προσπάθεια έρευνας και ανάπτυξης και ε, Επίση, να χρησιμοποιήσουμε τους σπόρους ε, για την προώθηση της έρευνα και τη ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο. Ένα άλλο τρόπος, ε, μια άλλη ρεαλιστική προσέγγιση για το θέμα θα μπορούσε να είναι να σκεφτούμε τι μπορούμε να καταστήσουμε υποχρεωτικό, δεσμευτικό σε μια νέα συνθήκη και τι θα μπορούσαμε να αφήσουμε στην ευχέρεια των κρατών, να προβούμε σε πολιτικές εταιρικέ σχέσεις μέσα στο πλαίσιο της Ένωσης, αλλά και με ε, άλλους εταίρους εκτός Ένωσης. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες και πιστεύουμε πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αν δούμε δηλαδή την μέθοδο Σέγγεν, όπου λειτουργήσε πολύ καλά. Ε, θα μπορούσε να είναι μια συμβιβαστική επιλογή που θα μας επέτρεπε να επιτύχουμε πρόοδο σε κάποια από τα στοιχεία αλλά όχι σε όλα τα στοιχεία που εξετάσαμε. Για να τα πετύχουμε όλα θα χρειαζόταν μια νέα συνθήκη. Και έρχομαι σε αυτό που εμείς θεωρούμε καλύτερη λύση που θα ήταν μια νέα συνθήκη για την ενέργεια, μάλλον μια νέα κοινότητα ενέργειας. Πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν το πιο αποτελεσματικό και καλύτερος τρόπος ε, μέσω της Ευρωπαϊκής Μεθόδου για να υπάρξουν δράσεις για όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρουμε στην έκθεσή μας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να, να κοιτάξουμε τα προηγούμενα του παρελθόντος και να έχουμε opt-in και opt-out, να επιτρέπουμε να είναι ανοιχτοί σε όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να τους δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν ή όχι opt-in ή opt-out. Μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε αυτή την προσέγγιση. Όπως ακολουθούμε ε, συνήθως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να έχουμε υπερεθνική διοργάνωση και θα πρέπει, όπως τονίζεται και στην έκθεση επανειλημμένα, θα πρέπει να εξασφαλίζουμε το ότι οποιαδήποτε νέα συνθήκη δεν θα καταστρέφει όσα φτιάξαμε τα τελευταία 50-60 χρόνια, το αποκαλούμενο ακεί, το κεκτημένο. Όλων αυτών δεδομένων το να ετοιμάσουμε μια νέα συνθήκη, το να διαπραγματευτούμε μια νέα συνθήκη, αυτό είναι κάτι περίπλοκο, είναι χρονοβόρο και είχαμε και την υιοθέτηση συνθήκη συνθήκης της Αβώνας και τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε κουραστεί κάπως με τις συνθήκες, οπότε ίσως ήταν πολύ φιλόδοξο να εξετάσουμε το δεχόμενο μιας νέας συνθήκης στο εγγύς ε, μέλλον. Μάρκ, ήδη είπε η Λή ποια είναι η προτίμησή μας οι νομικοί προτιμούν τη νέα συνθήκη. Ε, νέα όμορφα νομικά μέσα για τους νομικούς είναι ό,τι καλύτερο. Όμως πρέπει να είμαστε αρκετά ρεαλιστές και θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι χρειάζονται ε, κάποια ενδιάμεσα μέσα πιο ρεαλιστικά πρέπει να ακολουθούν πρώτα. Και αυτά τα πραγματιστικά βήματα θα πρέπει να οδηγήσουν προς την ενεργειακή κοινότητα την ευρωπαϊκή. Τόσο αφορά τα βήματα, θεωρούμε ότι το πρότυπο Σέγγεν προσφέρει τις καλύτερες δυνατότητες αυτού του τύπου. Θα πρέπει να ετοιμάσουμε έναν οδικό χάρτη, ένα πρόγραμμα και τα κράτη-μέλη που θέλουν να προχωρήσουν θα συμφωνήσουν επί των βημάτων και μετά θα αποφασίσουν για το επόμενο βήμα. Και όλο αυτό μπορεί να διαδοθεί σε όλη την Ευρώπη για διάφορα κράτη-μέλη. Μπορεί να έχει κανείς πολλές ομάδες και όχι μία ομάδα που θα κινούνται όλες οι ομάδες προς τον ίδιο στόχο. Και τελικό στόχος βεβαίως θα είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική. Στην έκθεση εντοπίσαμε κάποια παραδείγματα των συμφωνιών τύπου Σέγγεν που θα μπορούσαν οι πολιτικοί θα μπορούσαν να εξετάσουν και έχουμε και το ενεργειακό δίκτυο που είναι μία από τις λύσεις που μάλιστα είναι και σημαντική. Θα εξηγήσουμε γιατί. Η έκθεση εξηγεί πράγματι ότι ένα ενεργειακό δίκτυο που θα μπορούσε να έχει τη μορφή μια συνθήκη ενεργειακού δικτύου είναι ένα από, του βασικού τους βασικούς οικοδομικούς λίθους της αγορά. αυτής ενεργειακής αγοράς. Είδαμε ότι ας πούμε με ηλιακού ιστοριστέ μπορούμε να λειτουργήσουμε, να κινηθούμε καλύτερα στην Ισπανία από ό,τι στη Σκωτία. Έχουμε περισσότερους ανέμους όμως στο βορρά. Ενώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον ήλιο οι χώρε του Νότου άνεμο στο βορρά, ήλιο στο νότο. Και μπορεί να γίνει αυτή η συμβολή μέσω ενός υπερδικτύου, τεραστίου δικτύου που μπορεί να συναθρίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Ήδη έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον προηγούμενο για περαιτέρω συνεργασία όχι μόνο μεταξύ κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και με, με γείτονες είναι η συνθήκη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην ενεργειακή συνεργασία που εκεί υπάρχει εκτεταμένη συνεργασία όσον αφορά τα δίκτυα και όσον αφορά τους αναγκαίου κανόνες και ρυθμίσεις ώστε να λειτουργούν τα δίκτυα σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό θα συνεπάγεται και πολύ καλύτερο συντονισμό από ό,τι μέχρι τώρα μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Θα έχουμε τη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ενέργειας, την Acer, που θα ξεκινήσει από Μάρτιο του 2011 τις εργασίες της και αυτό είναι κάτι που θα διευκολύνει περαιτέρω το συντονισμό, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο και θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα. Υψηλότερο επίπεδο ολοκληρώσεως μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ανεξαρτήτων εκτελεστικών φορέων σε περιφερειακό και ακόμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα ασχολείται με καθήκοντα τύπου δικτύου. Ναι, αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός μοντέλου τύπου Σέγγεν, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλο, όσον ένα ενεργειακό ταμείο, αν θέλετε, που θα μπορεί να συντονίζει και να χρηματοδοτεί ανάπτυξη και έρευνα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η νέα προγράμματα, κάτι που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν από μόνα τους τα κράτη-μέλη. Αυτό δημιουργεί το πρόβλημα των πόρων και λείπουν τα χρήματα σήμερα και γι' αυτό στην έκθεσή μας θεωρούμε ότι αυτή η νέα συνθήκη, αυτό το νέο ενεργειακό ταμείο θα πρέπει να χρηματοδοτείται από άμεσους πόρους και όχι από εθνικά κονδύλια. Και ένα τέτοιο ταμείο θα μπορεί να από συνεισφορές εκείνων ή από ε, τέλη συμφορήσεως ή όταν πολλούνται διάφορα πιστοποιητικά ανταλλαγή ε, ρήπων ETS. Υπάρχουν κάποια προηγούμενα που μας δίνουν μια νομική βάση για ένα τέτοιο ταμείο. Αυτό είναι το δεύτερο μοντέλο και όπως είπε ήδη ο πρόεδρος Μπούζεκ εξετάσαμε και τον δεχόμενο συνεργασίας όσον αφορά την αγορά φυσικού αερίου ε, στο επίπεδο των διεθνών αγορών. Νομίζουμε ότι και αυτό είναι ένας τομέας όπου θα μπορούσε κανείς να εξετάσει τον δεχόμενο μιας ολιστικής συνεργασίας όπου δεν θα αποφεύγεται η σύναψη μακροπρόθεσμα με συνεργειακή συνθήκη αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να τα αποκριθούμε σε, άμεσα σε προκλήσεις αυτή που αντιμετωπίζουμε εμείς όπως είπε ο πρόεδρος Πούσεκ όπου τα κράτη-μέλη ανταγωνίζονται το ένα το άλλο για να υπογράψουν συμφωνίες με εξωτερικούς προμηθευτές και βλέπουμε μια διάδοση πολλαπλασιασμού πέτρελαγωγών στα βόρεια, στα νότια, ανατολικά και δυτικά και όλοι οι πετρελαγωγοί ανταγωνίζονται για περιορισμένους πόρους. Μια λύση πιο ορθολογική για μια πολιτική λογική θα είναι να δημιουργήσουμε ομάδες αγοράς φυσικού αερίου, σεβόμενοι πάντες όμως τους κανόνες των συνθήκων, κυρίως τους κανόνες περί ανταγωνισμού. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και η σύστασή μας δεν θέλει να αντιταχθεί στους ισχύοντες κανόνες των συνθήκων. Και καταλήγουμε στα συμπεράσματά μας. Η μελέτη μας ε, καταγράφει τις υφιστάμενες πολιτικές, προσφέρει ιδέες επιλογές. Όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν αν θεωρηθεί λογικό από πλευρά πολιτική. Αυτό είναι δικό σας θέμα βεβαίως και όχι δικό μας. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να σας δώσουμε μια ιδέα για μια ευρωπαϊκή ενεργική πολιτική, ποια θα έπρεπε να είναι, ποιες επιλογές θα οδηγήσουν σε μια τέτοια ευρωπαϊκή ενεργική πολιτική, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος Μπούζεκ. Μια ευρωπαϊκή ενεργειακή κοινότητα. Η ενεργειακή πλευρά πτυχή της ενώσεως. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους δύο προέδρους που μας προσεκάλεσαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένουμε να ακούσουμε τις ερωτήσεις σας Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Ήταν άκρως ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα ο συμπρόεδρος της συνεδριάσεως, ο κ. Φρανσίσκο Χαβιέ, Ρόχο Γκαρσία, να, να προεδρεύσει το επομένο τμήματος της συνεδριάσεως μας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ας ευχαριστήσουμε για τις εισηγήσεις της καθηγήτριας και του καθηγητή Φαντεβόλτε που ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και περνάμε στη συνέχεια θα σας διαβάσω τη σειρά που θα έχουμε για τις παρεμβάσεις απόψε. Όπως ξέρετε οι βουλευτές που θέλουν να παρεύουν πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο για ότι ζητούν τον λόγο. Έχει διανεμηθεί σε όλες τις αντιπροσωπείες. Γνωρίζετε λοιπόν πώς θα ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Θα δώσουμε τον λόγο όταν θα γνωρίζουμε τα ονόματα και στους ευρωβουλευτές και στους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων για τρία λεπτά κάθε παρέμβαση. Και έτσι το ίδιο η ίδια διαδικασία με την μπλε κάρτα για επερώτηση για 30 δευτερόλεπτα για ερωτήσεις σε σχέση με τους εισηγητές που παρενέβησαν πιο πριν. Μετά από αυτή την επεξήγηση περνάμε λοιπόν... Διακόπτει ο Πρόεδρος. Έχει τον λόγο. Εσείς κύριε έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα που συζητάμε, Κύριοι βουλευτέ, ε, εκπρόσωποι του Εθνικού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, όπω το συζητήσαμε το θέμα εδώ, η ενέργεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα τη Ευρώπη. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα μια οικονομική ύφεση. Μια απειλή όσον αφορά την εξάντληση των πόρων και απειλεί λόγω της αλλαγής του κλίματος. Και είναι δύσκολες στιγμές αυτές που περνά η Ευρώπη και η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις. Αυτές στιγμές κρίσης είναι όμως ταυτόχρονα και στιγμές μεγάλων ευκαιριών. Η ανάπτυξη ανανεωσίμων πηγών ενέργειας, η πράσινη ενέργεια, όλα αυτά μπορεί να είναι το κλειδί για μια νέα βιομηχανία που θα βασίζεται στην βιώσιμη ανάπτυξη και στις νέες τεχνολογίες οι οποίες θα μπορούσαν να μας δώσουν καλύτερη θέση στη διεθνή αγορά όταν βγούμε από την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να ρυθμίσει τον ενεργειακό τομέα, προσπάθησε να δημιουργήσει μια εσωτερική αγορά ενέργειας και προσπάθησε επίσης να καταπολεμήσει την αλλαγή του κλίματος. Παρ' όλα αυτά, οι εθνικές λύσεις που υιοθετήθηκαν από κάποια κράτη-μέλη, ή πιο μεγάλα ή πιο μικρά κράτη, είχαν αρνητικά αποτελέσματα. Παρενόχλησαν όσον αφορά την επίτευξη των δεθέτων στόχων και δημιούργησαν δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Για 30 δευτερόλεπτα έχετε το λόγο. Πολύ καλά. Θα ήθελα να σας πω, όπως είπε και ο κύριος Μπούζεκ, ότι συμφωνώ και εγώ με τα μέτρα αυτά που θα πρέπει να ληφθούν για να δημιουργηθεί αυτή η ευρωπαϊκή αγορά και αυτή η ευρωπαϊκή κοινότητα της ενέργειας. Έχω πολλά πράγματα να πω, αλλά νομίζω ότι έχω δυνατότητα να το κάνω κατά τη διάρκεια των εργασιών μας. Ευχαριστώ. Um, uh, oh, oh, uh, λοιπόν, τα σχόλιά σας τα δεχόμαστε πολύ ευχαρίστως, σας σήμεθα ευγνώμονες. Ταιριάζουν με τις απόψεις μας οι εθνικές λύσεις στα κοινά προβλήματα. Δεν είναι προφανώς αρκετά, αρκετές. Εστιαστήκατε στην αγορά σε αυτά που είπατε, στις δυνάμεις της αγοράς. Στην έκθεσή μας πιστεύουμε ότι οι δυνάμεις της αγοράς είναι κάτι που πρέπει να το υποστηρίξουμε διότι αυτές θα δώσουν τα αποτελέσματα στο τέλος. Όμως κάπως θα πρέπει να ελεγχθούν αυτές οι δυνάμεις. Και πώς να το πω. Ίσως πρέπει μια πιο κατευθυντική κατεύθυνση να δοθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων, πιο ελεγχόμενη κεντρικά ελεγχόμενοι. κάτι στην ανάγκη να αποφευθούν συγκρούσεις. Υπάρχουν χρήσιμα παραδείγματα που βλέπουμε στην πράξη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πεντελογωγό Ναμπούκο διάφορες χώρες συζητούν όχι μόνο με τις Ευρωπαϊκή Ενώσει, αλλά και υποψήφιε χώρες συμμετέχουν συνομιλίε, προσπαθώντα να πετύχουμε μια καλή λύση, μια αποδεκτή λύση αντί να περιμένουμε μέχρι ότου δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και να λύσουμε κάποια σύγκρουση πρόβλημα τέτοιο. Η προσέγγιση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι αποφυγή συγκρούσεων και η ενθάρρυνση της συνεργασίας. Υποστηρίζω τα όσα είπατε με άλλα λόγια. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι ότι όποιος θέλει να παρέμβει μέσα σε αυτά τα τρία λεπτά. Θα πρέπει να εγγραφεί εκείνοι που θέλουν να το κάνουν με την μπλε κάρτα να ξέρουν ότι θα έχουν 30 δευτερόλεπτα και μετά θα αφαιρείτε το μικρόφωνο. Θα λάβει τον λόγο ο κύριος Πατήτης παρακαλώ. Thank you, the President. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της συνεδρίασης. Πραγματικά συνενώνονται οι Ευρωπαίοι σήμερα για να συζητήσουν τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τους ενεργειακούς σκοπούς. Θα ήθελα να υπενθυμίσω το σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη σφαιρική διαδικασία και τις μεγάλες προσπάθειες του Προέδρου Μπούσεκ της Ευρωβουλής που με σθένος και κάθε προσπάθεια προσπαθεί να δημιουργήσει αυτή την ευρωπαϊκή κοινότητα. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ισπανική Προεδρία για την προθυμία για συνεργασία. Είναι μεγάλη πρόκληση για μας συνολικά στο μέλλον να μπορέσουμε σωστά να υλοποιήσουμε τις δράσεις μας για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Προσβλέπω σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις απόψε σε, αυτή, σε αυτόν τον κύκλο και ελπίζω ότι η έκβαση της συζήτησης δεν θα οδηγήσει σε δημιουργία μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Θα περάσουμε στη συνέχεια και θα λάβει τον λόγο η εκπρόσωπος της Ιταλικής Βουλής. Η κυρία Μαστρομάουρο, παρακαλώ, θα λάβει τον λόγο λεπτά. Πάνω απ' όλα θέλω να εκφράσω τι ευχαριστίε μου από πλευρά τη ε, Βουλή μα για την διοργάνωση αυτή τη συνεδριάσεω που δείχνει ξεκάθαρα πόσο βασικό είναι το θέμα τη ενέργεια ε, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την επίγνωση του στρατηγικού ρόλου που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπομειστεί όσον αφορά αυτό το θέμα. Η προοδευτική διεύρυνση τη πρόσβαση στην ενέργεια όσον αφορά τι αναδυόμενε χώρε και η μείωση τη ενεργειακή φτώχεια που είναι ένα φαινόμενο κάτι θετικό αυτό καθ' αυτό, μας οδηγεί σε μια αύξηση όμως του ανταγωνισμού όσον αφορά ε, την χρήση των ενεργειακών πηγών και καθορίζει αύξηση, δημιουργεί αύξηση πίεση όσον αφορά τα οικοσυστήματα και το κλίμα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση που εξαρτάται κατά σημαντικό τρόπο από τις εισαγωγές από περιορισμένε χώρε, αυτό το φαινόμενο μπορεί να έχει σημαντικέ συνέπειε όσον αφορά τον ασφαλή φοδιασμό ενέργεια, πέρα από την περιβαλλοντική πολιτική και πιο συγκεκριμένα για την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο. Η κρίση μεταξύ Ουκρανία και Ρωσία του φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια κατέδειξε σαφώ το πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη όσον αφορά τον εφοδιασμό τον ενεργειακό. Αυτή η κρίση ε, οδήγησε τα, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν τι πρωτοβουλίε θα πρέπει να αναλυφθούν για να εξασφαλιστεί συνέχεια και ασφάλεια εφοδιασμού ενέργεια σε βιώσιμε τιμέ. Και γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πρέπει να υπάρχει ποικιλομορφία στον από τι πηγέ και του προμηθευτέ και τι διόδου για τον εφοδιασμό σε ενέργεια. Είναι θεμελιώδη σημασία σε αυτό. Όπω και η εξοικονόμηση ενέργεια, η έρευνα και η καινοτομία, η τεχνολογική είναι στοιχεία βασικά για να μειωθεί η εξάρτηση από το εξωτερικά και ταυτόχρονα να μειωθεί η εκπομπή των αριθμών και πιο λεπτομερό πιστεύουμε ότι πέρα από τα συγκεκριμένα ε, συμφέροντα κάθε χώρα που ποικίλουν, ε, αν υπάρχει καλύτερο συντονισμό από πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεω, θα και για να πετύχουμε αυτό θα πρέπει να βελτιωθούν τα μέσα ε, αλληλεγγύης όσον αφορά την κρίση και για τον εφοδιασμό εισάγοντας διάφορους μηχανισμούς που θα αποφύγουν τη δημιουργία μπλοκαρίσματος στον αφορά τον εφοδιασμό ενέργειας. Θα πρέπει περισσότεροι πόροι να διατίθενται για να, πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση να χορηγούνται και να χρησιμοποιούνται όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις χρηματοδοτήσεις Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να εφαρμοστούν μέσα τα οποία θα βελτιώνουν την προσφορά ενέργειας και θα πρέπει να εφαρμόζονται περισσότερα μέτρα όσον αφορά το πακέτο κλίμα και ενέργεια και να δίνονται περισσότερα κίνητρα για να επιτυχάνονται οι στόχοι που έχουν αποφασιστεί όσον αφορά την εξοικονόμηση τη ενέργεια και πάνω απ' όλα για να δοθούν κίνητρα στην χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργεια που επηρεάζουν λιγότερο το περιβάλλον και τέλο θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί κοινή στρατηγική όσον αφορά τι σχέσει με τι χώρε προμηθευτέ. Όπω βλέπουμε, πρόκειται περί φιλοδόξων προκλήσεων και ταυτόχρονα είναι κάτι αναπόφευκτο για να εγγυηθούμε ένα σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το διεθνέ προσκήνιο τα επόμενα χρόνια που θα επηρεάζονται όλο και περισσότερο από την αυξανόμενη ρόλη αυτή, από την αυξανόμενη εξάρτηση και απέτηση ενέργειας. Πρόεδρο, πρόεδρος σας ευχαριστώ κυρία. Θα ήθελα να σας πω ότι θα δώσουμε προτεραιότητα σε εκείνους που έχουν εγγραφεί και όταν θα έχουν παρέμβει θα, λάβουμε, θα περάσουμε σε ερωτήσεις. Έχει τον λόγο το μέλος από την Γαλλική Βουλή, Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Λέγε για παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Oui, Αγαπητοί συνάδελφοι, οι προκλήσεις της ενεργειακής καταστάσεως είναι πολύ σημαντικές και γι' αυτό επικροτώ πλήρη την πρωτοβουλία σας κύριε Μπούζεκ. Είναι σημαντικά αλλά δεν τα συζητάμε επαρκώς και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα ακόμη δεν αρκούν αντιθέτως διότι από τη δεκαετία του 2000 υπήρχαν, υπήρχε μια στάθεια στην τιμή του ε, ενεργειακή, ε, διακοπές ενεργειακής παροχής ε, και όλα αυτά επηρέασαν την Ευρώπη η οποία εισάγει 100% του πετρελαίου και 60% του φυσικού αερίου και αυτά τα στοιχεία θα είναι πιο σημαντικά στο μέλλον. Άρα οι κλιματολογικές αλλαγές ζητούν να μειώσουμε την ε, το διοξίδιο του άνθρακος άρα ε, χρειάζεται μία διαφοροποίηση των πηγών ιδίως για το αέριο πρέπει να αναφερθούμε στον αγωγό αερίου προς την, τους αγωγούς αερίου προς την Ευρώπη Nord Stream, Strauss Stream, Nabucco και την παροχή μεθανίου θα πρέπει τα δίκτυα αυτά να συμπράξουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων τα κράτη θα πρέπει ε, να μπορούν να διαλέγουν σύμφωνα με τις επιταγές συνθήκης της Λισαγώνας ε, τις ενεργειακές πηγές που επιθυμούν αλλά συγχρόνως να δεσμευτούν ότι θα μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος που είναι ένα θέμα που μας ε, αφορά όλους. Μία άλλη άποψη αναφέρεται στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες, να υπάρχει δηλαδή μία ενεργειακή διπλωματία όπως ελέγχθη προηγουμένως. Όπως απέδειξε η κρίση του αερίου του 2009, τον Ιανουάριο 2009, χρειάζονται αλλαγές. Δηλαδή, εγώ που είμαι πρόεδρος της Γαλλικής Βουλής, ε, μπορώ να σας πω ότι έχουμε ενισχύσει την ε, ε, απόφαση ε, η οποία ελήφθη για να προωθηθεί η αλληλεγγύη μεταξύ κρατών, να υπάρξει περισσότερη χρηματοδότηση, να υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το πακέτο των υποδομών που έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά μία νέα συνθήκη που αναφέρθηκε προηγουμένως είμαι αντίθετος. Είχα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εθνοσυνέλευση, είδα τι προβλήματα δημιουργεί η εκπόνηση ενός τέτοιου εγχειρήματο. Θα χρειαστεί λοιπόν μία καλύτερη συνεργασία και μία πολιτική θέληση ισχυρή. Αυτό είναι η προϋπόθεση για να επιτύχει μία πραγματική ενεργειακή πολιτική. Και πάλι ε, συμφωνώ με την πρωτοβουλία των κυρίων ε, Μπούζεκ και Ντελόρ. Σας ευχαριστούμε κύριε στη συνέχεια. Ο κύριος Ευρωβουλευτής Ρώση, παρακαλώ, θα λάβει τον λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, σα ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο για να συζητήσουμε την ενέργεια στον 21ο αιώνα. Θα πρέπει ωστόσο να ξεκινήσω με μια επίκριση, γιατί τα επίσημα κείμενα διανέμονται μόνο σε ορισμένε γλώσσε, και παράδειγμα λείπουν τα Ιταλικά. Και γι' αυτό θα πρέπει να πω, Πρόεδρε, ότι είμαι πολύ δυσαρεστημένο. Να περάσω στο επιχείρημα τώρα για το οποίο βρισκόμαστε εδώ σίγουρα, δεν υπάρχουν αμφιβολίε. πρέπει να βρεθεί κοινή ενεργειακή πολιτική για την εξασφάλιση των εφοδιασμού για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και για να προσφέρεται μια υπηρεσία σε μια ε, λογική και εγγυημένη τιμή σε ολόκληρη την Ένωση. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, διαρκώς αυξημένο κόστος για τις, τις διάφορες πηγές ενέργειας. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ε, αθέμητο ανταγωνισμό ανάμεσα στις διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε διαφορετικές πραγματικότητες. Άρα λοιπόν το να έχουμε να κάνουμε σε κοινοτικό επίπεδο με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο σημαίνει ότι θα έχουμε και καλύτερες τιμές. Πρέπει επίσης να επενδύσουμε στην έρευνα για να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι πράσινες πηγές θα πρέπει και εκεί να μας βρουν ενωμένου. Ε, αφού η κάθε χώρα, μάλλον όσο η κάθε χώρα θα ταξιδεύει μόνη της με διαφορετική ταχύτητα δεν θα έχουμε ωφέλ για τους πολίτες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελλείψη στον αγώνα κατά της περιορισμού των εκπομπών είναι αγώνας τρίτων χωρών όπως η Ινδία, η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής. Ίσως θα πρέπει να επιβάλλουμε φόρους ε, στα εμπορεύματα τρίτων χωρών που δεν δεσμεύονται για το περιβάλλον. Μια Ένα πραγματικό φόρο για το διοξείδιο του άνθρακα που θα τηρεί το ρητό ο ρηπαίνων πληρώνει. Δεν μπορούμε μόνο να συζητάμε με το, για το κλίμα και το περιβάλλον όπως με τους 15 στην Κοπενχάγη και όπου λόγω υπερβολικού ζήλου η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε ένα έγγραφο το οποίο εγώ αποκάλεσα ως ε, τη βίβλο των ε, ονείρων που τελικά όμως κατέληξε σε μια αποτυχία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το νέο βάρο που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χάρη στη συνθήκη τη Λισαβόνα, να υποβάλουμε προτάσεις και αιτήματα σοβαρά, αξιόπιστα, που ολόκληρο ο κόσμο ε, ε, ο εργαζόμενο θα οφείλει και θα μπορεί να δεχτεί. Σε μια περίοδο τέτοια ε, παγκόσμια ύφεση την οποία διανύουμε, το να προχωρούμε χωριστά δεν θα μας οδηγήσει τίποτα συγκεκριμένο. Θα σας ε, εκφράσω μια δική μου σκέψη, πρόεδρε, αγαπητέ πρόεδρε Μπούζε. Και εσείς υποβάλλατε ένα έγγραφο για την ανενέργεια, ένα έγγραφο το οποίο εγώ εκτίμησα και σας το είπα. Θα σας καλέσω να συνεργαστείτε με όλους ώστε ένα τέτοιο, αυτό το κείμενο διευρυμένο να αποτελέσει τη βάση για τις προτάσεις της του δικού μας κοινοβουλίου στην ε, επόμενη ΚΟΠ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε. Στη συνέχεια, ο κύριος ε, Γερουσιαστής από την Πολωνία παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλο τεράστιο ενδιαφέρον παρακολούθησα τις παρεμβάσεις των φιλοξενουμένων και συμφωνώ απόλυτα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εθνικές ενεργειακές πολιτικές και όπω όπως ακούσαμε από τον πρόεδρο της Ευρωβουλής Γιέζη Μπούζεκ, αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι μια ενιαία κοινή κοινοτική στρατηγική για τα ενεργειακά θέματα. Στο παρελθόν καταδείχθηκε ότι τα προβλήματα ασφάλειας της κάλυψης ε, των ενεργειακών αναγκών δεν είναι μόνο θέματα των ΜΜΕ αλλά απειλούν την επιβίωσή μας. Κάποιες χώρες έκαναν μεγάλες προσπάθειες, η Πολωνία για παράδειγμα, να βρουν λύσεις με βάση την αρχή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Όμως η συνολική κατάσταση δεν βελτιώθηκε. Αυτή επίσης είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εφιστά την προσοχή σε κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες χωλένουν με βραδύ ρυθμό όσον αφορά την υλοποίησή τους, ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα υποδομών, ενεργειακών υποδομών. Εμείς θεωρούμε ότι σε μια ενωμένη Ευρώπη χρειαζόμαστε άμεσα αποτελεσματικές αποφάσεις και διαδικασία λήψεων αποφάσεων που θα διασφαλίζουν μια ενιαία κοινοτική αγορά ενεργειακών πόρων, ώστε να είναι δυνατόν να έχουμε πρόσβαση σε ενεργειακά προϊόντα σε προσιτές τιμές, ώστε από τα λόγια να περάσει η Ευρώπη στις πράξεις. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια διακήρυξη Μία διακήρυξη, για παράδειγμα, στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι και ποιοι θα είναι οι χαμένοι από αυτήν την κοινή ενεργειακή πολιτική μας. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία, πιστεύω, με μια τέτοια τοποθέτηση, χώρες θα μπορέσουν να κινητοποιηθούν και να αναδυθούν από αυτή την κρίση με μεγαλύτερη επιτυχία και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους με μεγαλύτερη επιτυχία. Οι πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την Πολωνία και άλλες χώρες κατέδειξαν ότι η ασφάλεια κάλυψης των ενεργειακών αναγκών δεν είναι μόνο η μείωση όσον αφορά την εξάρτησή μας από πετρελαγωγούς και αγωγούς φυσικών αερίων αλλά είναι η διασφάλιση της, ε, των ενεργειακών αναγκών μας ε, όταν για παράδειγμα τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας ε, για τον ένα ή άλλο λόγο πλήττονται ή καταστρέφονται έστω εν μέρη και υφίστανται ζημιές και αυτό φυσικά αναπόφευκτα οδηγεί σε ε, υψηλότερο κόστος, σε μεγαλύτερες δαπάνες. Συμφωνώ στις ε, δυνατές ε, κατευθύνσεις δράσης που σκιαγράφησε ο πρόεδρος Μπούζεκ και όσον αφορά τις προκλήσεις, είναι παγκόσμιες οι προκλήσεις αυτές και απαιτούν, ζητούν από εμάς ε, ενιαίες ε, ε, σφαιρικές απαντήσεις. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε σε περιφερειακό επίπεδο να υλοποιήσουμε. Θεωρώ ότι η χάρτα υποχρεώσεων και καθηκόντων είναι μια νέα ευκαιρία. Πρόεδρος, περνάμε στη συνέχεια και θα δώσουμε τον λόγο στον κύριο εκπρόσωπο από τη Λιθουανία παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα δρατώμενος της ευκαιρίας το σχέδιο που προτάθηκε για την δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας στην Ευρώπη να το χαιρετήσω. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε πολυμορφοποιημένες υποδομές και να ε, πολυμορφοποιήσουμε τις, ε, την εξάρτησή μας από ενεργειακούς πόρους. Η λιθουανική στρατηγική όσον αφορά τα θέματα ενέργειας βασίζεται στη συνεργασία και στην ασφάλεια. Είμαστε και εμείς ε, ως Λιθουανοί υπέρ της δημιουργίας ενός ενεργειακού δικτύου στην περιοχή της Βαλτικής. Ε, αυτό θα οδηγούσε και θα διασφάλιζε την ενεργειακή ολοκλήρωση και με βάση την περιφερειακή ολοκλήρωση αυτό που προσπαθούμε ως Λιθουανοί είναι να δημιουργήσουμε εμείς ένα κομβικό σημείο, ένα σταυροδρόμι μεταξύ των ε, ανατολικών χωρών και των σκανδιναβικών χωρών και έτσι να υπάρξει η πιο αποτελεσματική διαμόρφωση των ροών. Η δημιουργία της ενεργειακής αυτής κοινότητας θα συνεισφέρει η αλληλεγγύη να διασφαλιστεί όπως ε, στη συνθήκη της Λισαβόνας κατοχυρώνεται Ελπίζω ότι η ενεργειακή ασφάλεια θα είναι ένα θέμα το οποίο θα είναι ανοιχτό, να είναι, θα είναι προσβάσιμο, προσπελάσιμο σε όλα τα κράτη που θα θέλουν να συνεργαστούν. Και έτσι από πλευράς Λιθουανικού Κοινοβουλίου το ενεργειακό πρόγραμμα, το σχέδιο αυτό θα το συζητήσουμε. έχω βεβαιότητα ότι η Λιθουανία θα είναι μεταξύ των χωρών που θα οικοδομήσουν την ενεργειακή κοινότητα. Πρόεδρος, εξ ονόματος της ε, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής θα λάβετε εσείς τον λόγο παρακαλώ. Uh, uh, uh, Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα το ότι η ε, Κοινωνική και ε, Οικονομική Επιτροπή προσκλήθηκε να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση. Και όπως ίσως πιθανόν γνωρίζετε, έχουμε πολυάριθμες γνωμοδοτήσεις που εγκρίναμε για τα προβλήματα τα οποία έχουν τεθεί υπό συζήτηση ε, εδώ σήμερα. Θα ήθελα να αναφερθώ στην τελευταία μας γνωμοδότηση και σε αυτήν ε, να αναφερθώ, διότι αυτή ταιριάζει με το θέμα το οποίο συζητάμε. Είναι αυτό το οποίο αφορά το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική ανάπτυξη όσον αφορά τεχνολογίες χαμηλού, χαμηλών εκπομπών άνθρακα, χαμηλών εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα. Αναφέρθηκε ότι αυτό θα είναι το κλειδί για την επίλυση των προβλημάτων, για την αηφορία και την ανταγωνιστική διασφάλιση των ενεργειακών πόρων της Ευρώπης. Όπως αυτό μπορεί όμως ε, με τεράστιες κοινέ προσπάθειες, κοινοτικέ προσπάθειες να επιτευχθεί. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο συζητάμε εδώ. Πόσο κοινοτικέ πρέπει να είναι οι διαδικασίες μας, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ανησυχεί βαθύτατα όμως διότι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη και προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις τα κονδύλια τα οποία θα απαιτηθούν υποεκτιμούνται και γι' αυτό είναι κατεπήγον ώστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη και από την ιδιωτική οικονομία και τις επιχειρήσεις να υπάρξει ένα, ε, ένα πιο διευρυμένο οικονομικό πρόγραμμα, ένα οικονομικό σχέδιο το οποίο θα ε, δραστηριοποιήσουμε και να έχουμε υπόψη και τις, τα πιστοποιητικά εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα καθώς επίσης και την εισαγωγή ενός τέλους για τον άνθρακα, ενός φόρου για τον άνθρακα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο για την προστασία του περιβάλλοντος ε, θα αντληθούν ε, κονδύλια από την ευρωπαϊκή οικονομία. Θα ήταν παράλογο να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια για άλλους σκοπούς ε, αντί να χρησιμοποιηθούν για τις εξειδικευμένες τεχνολογίες που θα πρέπει να μπορέσουν να αναπτυχθούν σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Είναι η πιο σαφή τοποθέτηση αυτής της γνωμοδότησής μας και θα ήθελα να περάσω τώρα στα αγγλικά στην παρέμβασή μου για να αναφερθώ σε ένα παράθεμα, σε μια πρόταση που ε, σε σχέση με τη γνωμοδότηση Affordable Energy, προσιτή ενέργεια, που θα είναι το αίμα, η, η δύναμη της οικονομίας μας. Γνωρίζοντας σε σχέση με την πρωτοβουλία την οποία έχετε αναλάβει, είναι απόλυτα σαφές ότι μόνο με κοινέ προσπάθειες μπορούμε να πετύχουμε με αυτό το στόχο. Και το πρόβλημα δεν πρέπει να το υποτιμούμε με κανένα τρόπο. Τα επιμέρους κράτη-μέλη δεν θα είναι μόνα τους σε θέση να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα. Το αν θα είμαστε από κοινού σε θέση να το επιλύσουμε θα ε, μπορέσει να διασφαλιστεί μόνο να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κύριε. Στη συνέχεια ο κύριος ε, Γερουσιαστής από την Ιταλία παρακαλώ. Ναι, Ευχαριστώ. Τελευταία χρόνια η Ιταλία αύξησε τι προσπάθειε που κατέβαλε για τη με τι ενεργειακέ πολιτικέ που περιγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, προβαίνουμε στην υλοποίηση μια ενεργειακή αγορά πιο απελευθερωμένη που εξασφαλίζει μεγαλύτερο ανταγωνισμό με μείωση των τιμών των ενεργειακών ε, ηλεκτρική ενέργεια φυσικού αερίου, ανάπτυξη υποδομών στατικικών για τη μετάδοση ηλεκτρική ενέργεια και δημιουργία νέων συστημάτων αποθέματο αποθήκευση φυσικού αερίου και όπω και το πακέτο κλίμα και ενέργειας προωθούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ιταλία τα τελευταία χρόνια άνοιξε την αγορά της ηλεκτρική για σε διάφορους φορείς και βασίζεται στην απελευθέρωση του τομέα της φυσικού αερίου μέσω μιας γενναίας μεταρρύθμισης η οποία εξετάζεται τώρα από το τελικό κοινοβούλιο. Μια μεταρρύθμιση η οποία βασίζεται σε μεγαλύτερη συμμετοχή των μεγάλων καταναλωτών ενέργειας με προγράμματα υλοποίηση ε, νέων συστημάτων αποθήκης φυσικού αερίου και η Ιταλία θα μπορεί λοιπόν να αυξήσει τα αποθέματά της και να έχει μεγαλύτερη ε, ασφάλεια εφοδιασμού. Αυτά μπορεί να ωφελήσουν όλα τα κατημέλη διότι οι επενδύσει των επόμενων ετών όσον αφορά την αποθήκευση ενέργεια φυσικού αερίου θα επιτρέψει στην Ιταλία να είναι πραγματικό κόμβο φυσικού αερίου στη Μεσόγειο. Και όσον αφορά το τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η χώρα μου ξεκίνησε με την παρούσα κυβέρνηση μια προσπάθεια για μεγαλύτερη ποικιλομορφία όσον αφορά τις πηγές ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η ποικιλομορφία έχει τρία βασικά σημεία. Ε, την προώθηση των ανεωσίμων πηγών ενέργειας όπως ζητείται από το πακέτο 2020-2020, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς να ξαναρχίσει ε, ε, οι πυρηνικοί σταθμοί θα να, ε, θα δημιουργηθούν αμέσω συμφωνιών με τα κράτη-μέλη για την δημιουργία κατασκευών εγκαταστάσεων τρίτη γενιά. Στην πρώτη γραμμή από πλευρά τεχνολογία και ασφαλεία θα είναι αυτή η πυρηνική σταθμή. Και σε αυτή την περίπτωση η παραδρομολόγηση του πυρηνικού προγράμματο στην Ιταλία θα μα βοηθήσει να μειώσουμε σημαντικά το κόστο ηλεκτρική ενέργεια. Και δράτω με τι ευχέ που έχω αυτό το τελευταίο λεπτό στη θέση μου να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ την έκθεση των δύο νομικών και από τη δική μας πλευρά πιστεύουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Μυθιστικός Φορέας θα πρέπει να κινείται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο θα πρέπει να είναι το θέμα της διανομής εξασφάλισης του φωτιασμού ενέργειας και το δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να είναι κάτι με το οποίο ασχολείται η Ευρώπη για μια πολιτική παγκόσμια ενεργειακή με χαμηλή συνέπεια και επιπτώσει για το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις εταιρείε μας ε, υποπίεση οικονομική που οφείλεται στο μεγάλο κόστος των ελλακτικών πηγών ενέργειας που αν αυτό δεν συμμορφωθεί με τη διεθνή οικονομία θα, βάζει, θα βάλει την Ευρώπη εκτός ε, διεθνούς ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κύριε. Στη συνέχεια η γερουσία της Τσούσκοβα από την Τσεχία παρακαλώ. Έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα θα ήθελα να συμβάλλω στη συζήτηση αυτή από δύο σκοπιές. Καταρχήν η απάντηση της Ευρώπης ήταν αντίδραση στην έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να υπάρξει ειρήνη στην Ευρώπη και <clears throat> για να υπάρχει μία συνενετική χρήση των πόρων. Από εκεί ξεκίνησε η συνθήκη άνθρακος και χάλιβος. Τώρα όμως πολλοί θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι κάτι δεδομένο και πολλοί επανέρχονται σε εθνικιστικές τάσεις. Υπάρχουν όμως δύο τομείς στις οποίες χρειάζεται κοινοτική προσέγγιση. Καταρχήν ε, η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και τα θέματα της ασφαλείας διότι κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα μόνο του. Είναι τόσο προφανές ώστε θα έπρεπε να μπορεί κανείς να εξηγήσει ε, το θέμα αυτό σε κάθε Ευρωπαίο. Έχουν γίνει ήδη πολλά και αυτό το συνέδριο είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, προς την ίδια κατεύθυνση και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπούζεκ για αυτή την πρωτοβουλία. Θέλω όμως να θίξω και άλλο ένα θέμα, το οποίο εάν δεν επιληθεί δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Χρειαζόμαστε καλά επιμορφωμένα άτομα τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν την διαβίου μάθηση που μπορούν να έχουν την σωστή εκπαιδευτική και ηθική βάση διότι η ε, διαχείριση των ενεργειακών πόρων είναι πολύ σοβαρό θέμα. Υπάρχει μια τέτοια πολιτική στην Τσεχία αλλά όταν μιλάμε στην Ευρώπη για ασφάλεια ενέργειας και παροχής ενεργείας πρέπει να σκεφτούμε ποιοι θα τα εξασφαλίσουν για λογαριασμό μας και η εκπαίδευση και ε, η επιμόρφωση είναι θέμα για τα κράτη-μέλη αλλά αν η κοινή πολιτική είναι στρατηγική κοινοτική ε, τότε θα πρέπει η Ευρώπη να ενισχύσει τις εξελίξεις όχι μόνο στον τομέα της ενεργείας αλλά και της τεχνικής ε, ε, εκπαιδεύσεως, της κινητικότητας, της διαβίου μάθησης που θα πρέπει να αποτελέσουν την κορονίδα των επιτεύξεων της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούζεκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ομιλητή που προείδρευσε ε, σε αυτό το τμήμα της συζήτησης. Επανέρχομαι τώρα στην Προεδρία και έχουμε ακόμη 8 ομιλητές. Έχω εδώ έναν κατάλογο των ατόμων που έχουν ζητήσει το λόγο και θα ήθελα να περιοριστείτε σε σχόλια 2,5 λεπτών, δηλαδή 1,5 λεπτό λιγότερο από τους προηγούμενους ομιλητές. Επιμένω σε αυτό και ο επόμενος είναι ε, ε, πρόσωπος του Αγγλικού Ράιστακ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να ε, είμαστε παρόντες ε, και να συζητάμε αυτά τα σημαντικά θέματα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εξαιρετική ε, ε αυτό τον εξαιρετικό περίγυρο και τις παρεμβάσεις. στα ενεργειακά θέματα είναι όχι μόνο σημαντικά για να πετύχουμε μια καλύτερη συνεργασία, αλλά είναι σημαντικό να δούμε ποια, ποιοι ενεργειακοί πόροι θα πρέπει να επιλεγούν για αυτή τη συνεργασία. Χρειαζόμαστε καλή επιλογή στόχων ε, και μια σύμβαση συνθήκη για την ενέργεια που θα βασίζεται σε αηφορία και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς επίσης ως εναλλακτικέ δυνατότητες και την πυρηνική ενέργεια. Χρειαζόμαστε φυσικά ένα βελτιωμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Ακόμα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σημαντικό στοιχείο. Είναι μια πρόκληση για την ευρωπαϊκή οικονομία και δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης σε αυτόν τον τομέα. Μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Η αιωλική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η, η ενέργεια από υδάτινους πόρους είναι πόροι ενεργειακοί με τους οποίους θα είμαστε ανταγωνιστικοί και μπορεί η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική. Επιπλέον θεωρούμε ότι με βάση τα ανανεώσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν πολλές νέες θέσεις ε, ε, εργασίας να δημιουργηθούν. Επιπλέον αυτό είναι μια ενέργεια, ένα είδος ενεργειακού πόρου που σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μπορούν, μπορεί να αναπτυχθεί Ενδιαφερόμαστε λοιπόν άμεσα και ιδιαίτερα να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε αυτό το ενεργειακό μέτωπο με τις άλλες χώρες. Πρέπει να διαρωτηθούμε όμως τι επιθυμούμε και θα θέλαμε να έχουμε ένα στόχο στον οποίο θα επικεντρώνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ για αυτή την περιεκτική παρέμβασή σας στη συζήτηση. Ο κύριος Ρομπέρτο Τορτόλη, επόμενος από την Ιταλία. <clears throat> Ευχαριστώ η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έδειξε θάρρος όσον αφορά ε, τον πρωτοπόρο ρόλο που θέλει να δραματίσει όσον αφορά τις μελλοντικέ πηγές ενέργειας ε, και για την αντιμετώπιση των πνευμάτων του περιβάλλοντος. Το πακέτο ενέργεια και κλίμα δείχνει την επίγνωση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ανάγκη να αντιμετωπιστούν από κοινού τα δύο πτυχέ τη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τι συνέπειε που έχει η ενέργεια στο περιβάλλον όσον αφορά τι εκπομπέ τη ρηπαντικέ. Τι τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να βρει ένα προωθημένο σημείο ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα και τη προωθήσεω τη τεχνολογική προόδου και τη ενημέρωση των παραγωγικών διαδικασιών ε, και την προστασία του οικονομικού τη συστήματο που βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό ακόμα επί των δραστηριοτήτων των κατασκευαστικών. Δεν κατάφερε όμω η Ευρώπη να παίξει τον πλήρη ρόλο τη όσον αφορά τη διάσκεψη τη Κοπενχάγη και ίσω αυτό δεν είναι κακό, διότι αν από τη μια πλευρά είναι θεμελιώδε να προχωρήσει προχωρήσουν στην κατεύθυνση της μέγιστης προσοχής όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα. Την άλλη πλευρά δεν είναι σωστό να εστερνιστούμε τη θέση της αλλαγής του κλίματος όταν γίνεται μια συζήτηση σε επιστημονικό επίπεδο ε, αμφίσιμο όσον αφορά τη θέρμανση του πλανήτου και ότι οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παρετηθούμε από την επιδίωξη με συνέπεια μια στρατηγικής που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπομισθούν όλοι οι παντέ τι ευθύνε του, ξεκινώντα από τι πιο ανεπτυγμένε οικονομίε και να συνεχίσουμε με τι χώρε τι αναδυόμενε όπω αποκαλούνται. Αλλά θα πρέπει με ρεαλισμό πολιτικό να προχωρήσουμε και όχι με ιδεολογία πολιτική. Θα πρέπει επίμον η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει να κινηθεί στα διεθνή φόρα για να ζητήσει από όλου να επομιστούν τι ευθύνε του, αλλά δεν θα πρέπει να κάνει βήματα αδικαιολόγητα προ τα μπρο. πρόσφατη απόφαση να πάρει παρετηθούμε πάνω από 20 30% τη μείωση των εκπομπών ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτή τη λογική ε, και λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης της παρούσης που δεν επιτρέπει να υποστηρίξουμε το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η αλλαγή των παραγωγικών συστημάτων που θα έπρεπε να γίνει. Η ταυτόχρονη συρρήκνωση της ενεργειακής ζήτησης που προέρχεται από τη μείωση της παραγωγής δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει ε, σε μια σταθε... να θεωρήσουμε ότι υπάρχει σταθερή τάση. Θα αυξηθεί η ζήτηση ενέργειας τα επόμενα χρόνια πιστεύω και η μείωση της χρήσεως των ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να συνεχιστεί σε μείωση προς όφελος της πυρηνικής ενέργειας και των ανενωσίμων πηγών ενέργειας. Στην παρούσα κατάσταση όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών είναι βασικά σκόπιμο να κινηθούμε όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, όσον αφορά την ανάπτυξη πιο προθυμένων ενεργειών που έχουν μικρή συνέπεια για το περιβάλλον, όπως είναι ενώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια κυρίως ε, στον τομέα της ε, έρευνας. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε. Ο κ. Αντζεζίπ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ καλό το θέμα που τίθεται. Αυτή, αν θέλουμε να έχουμε ευρωπαϊκή ενεργική κοινότητα ή όχι. Και χαίρομαι που το συζητούμε εδώ με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο ε, ε μας οδήγησε σε πολύ σημαντικές ε, θεωρίες που ακούστηκαν, ενδιαφέρουσες θεωρίες από κάποιους ομιλητές. Ε, με ενδιαφέρον άκουσα το πώς οι ενεργειακές πολιτικές που προσπάθησαν να εφαρμόσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχαν λοιπόν πέρα από την επικύρωση της συνθήκης της ε, Λισαβόνας μιλούσαμε για το μέλλον της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που ήταν ένα από του λόγου ύπαρξη τη Λισαβόνα. Τώρα που έχουμε στη θήκη τη Λισαβόνα, φαίνεται ότι λησμονούμε ότι υπάρχει ανάγκη για μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Και από του λόγου για του οποίου θέλαμε τη συνθήκη τη Λισαβόνα, κυρίω στην χώρα μου, την Πολωνία. Δοθήσει τη οικονομική καταστάσεω που επικρατεί στην ε, Πολωνία. Των περιστάσεων που επικρατούν. Ε, συμφωνώ λοιπόν κατά πολύ με αυτά που είπε ο πρόεδρος Μπούζεκ για ο οποίος συνέβαλε στη διοργάνωση αυτής της συνεδριάσεως. Εκτιμώ και αυτά που μας είπαν και οι προσκεκλημένοι μας ομιλητές, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις νομικές πτυχές του ζητήματος που ζητούμε. Η ΕΚΑΧ, η Οικονομική Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, ήταν πιο επιτυχής από ότι η ενεργική πολιτική που ακολουθήσα μέχρι τώρα. Η ΕΚΑΧ τώρα έχει εκπνεύσει και όμως ε, δεν έχουμε κάτι καινούριο να αντικαταστήσει την ΕΚΑΧ εν μέρη λόγω της ε, που αντιμετωπίζαμε. Βλέπουμε μεγαλύτερο εθνικό εγωισμό να επικρατεί. Αρκεί κανείς να δει τη δουλειά που γίνεται όσον αφορά τον ασφαλή εφοδιασμό σε φυσικό αέριο στο μέλλον για να το καταλάβει αυτό. Είχαμε ομόφωνη άποψη στην Επιτροπή Βιομηχανίας και τώρα και τώρα λέω, βλέπουμε ότι διεξάγονται συζητήσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του θέματος αυτού και πιστεύω ότι μια ομόφωνη άποψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να έχει θετικές συνέπειες όσον αφορά τις απόψεις των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να απομακρυνθούν, πιστεύω, από τους εγωισμούς τους. Ε, Λένα Κολάτσκα Μπομπίνσκα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας ε, οι οποίοι... Ε, Ευχαριστώ όλους σας που συνεισφέρατε στην έκθεση και στη συζήτηση των συναφών θεμάτων και θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο Μπούζεκ για το ότι συγκάλεσε αυτή την σύνοδο, αυτή τη συνεδρία. Επίσης θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί όχι λόγω της κρίσης αλλά επειδή έχει μεγάλα προγράμματα και εγχειρήματα και μεγάλες ζωντανές ιδέες. Δεν πρέπει η κρίση να είναι η μας, ε, το μόνο μας κίνητρο. Είναι μια ιδέα που θα μπορούσε λοιπόν να μας βοηθήσει να κινητοποιήσουμε όλο το δυναμικό της Ευρώπης ε, και να κάνουμε κάτι. Κάπως ε, ανησυχώ πρέπει να πω για αναφορές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αυτή τη στιγμή κινείται προς τα πίσω, ο πισθοδρομίος όσον αφορά θέματα ενεργειακά. Αυτό είπαν αρκετοί και ο λόγος γι' αυτό είναι, πρέπει να πούμε, ότι τα κράτη-μέλη ακολουθούν διαφορετικά και σατραπούς διαφορετικές κατευθύνσεις και πορείες. Τίθεται το ερώτημα, τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, δεδομένου ότι τα εθνικά συμφέροντα μέχρι σήμερα δεν συνεισέφεραν στο να υιοθετήσουμε και να προαγάγουμε μια κοινή κοινοτική ενεργειακή πολιτική. Μέχρι σήμερα αποτύχαμε λοιπόν και είναι σαφές αυτό. Το ερώτημα τίθεται πώς μπορούμε να κινηθούμε από την φάση των ιδεών και των προτάσεων στην φάση της υλοποίηση και των πράξεων. Τι θεωρεί ο πρόεδρος Μπούσεκ ότι μπορεί να γίνει. Σας ευχαριστώ κύριο Τσάρλς Τάνοκ παρακαλώ. Θα λάβει τώρα τον λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινό. Um, Σας ευχαριστώ πρόεδρε Μπούσεκ για αυτή την πρωτοβουλία. Λυπούμε και θέλω να πω σε σχέση με την συνένεση ή την ομοφωνία δεν μπορώ να δω πολιτική βούληση να ε, επενδύεται σε ε, αυτή την ε, μεγάλη ιδέα. Είναι προτεραιότητα των κρατών μελών και στην ε, οικονομία της, ε, των χαμηλών εκπομπών ε, άνθρακα υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό. Η ομάδα μου έχει μια θα έλεγα μειονοτική θέση. Πιστεύουμε ότι σε σχέση με την, τα θέματα της διασφάλισης των ενεργειακών αναγκών μας θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε την δυνατότητα της ε, ε, ομοφωνίας και πρέπει να δούμε το πώς θα διαμορφωθούν όλα αυτά. Γενικά όμως εμείς ε, προτιμούμε την διακυβερνητική συνεργασία ως μια μελλοντική συνιστόσα χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της συνθήκης το 194 τους κανόνες της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και τους κανόνες για τον ανταγωνισμό. Δεν βλέπουμε την ανάγκη να υπάρχει μια νέα συνθήκη συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ενεργειακά θέματα που θα ε, υποκαταστήσει ε, αυτά τα θέματα. Εμείς ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο απορρίπτουμε μια οποιαδήποτε νέα συνθήκη, οποιαδήποτε νέα συνθήκη και δεν μπορούμε να δούμε πώς θα μπορούσε να εγκριθεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Η διευρυμένη συνεργασία θα μπορούσε να είναι μια δυνατότητα στην οποία θα μπορούσαν να εμπλακούν κράτη-μέλη και σε σχέση με το ότι την ρυθμιστική αρχή είναι και αυτό κάτι το οποίο εμείς θα απορρίπταμε. Καλύτερο είναι η συνεργασία μέσα στο πλαίσιο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Επίσης ε, έχουμε ε, προβληματικούς τομείς, ε, όμως όσον αφορά την δυνατότητα να δραστηριοποιηθούμε για την αγορά ενεργειακών πόρων όπως του φυσικού αερίου, είναι κάτι το οποίο εθελοντικά τα κράτη μελη θα μπορούν να αναλάβουν ως πρωτοβουλία και υποστηρίζουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Το ενεργειακό μείγμα το οποίο θα ε, ήθελε κανείς να ακολουθήσει σε σχέση με ένα ε, μέλλον διασφάλισης των ενεργειακών πόρων και όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια πρέπει να είναι θέμα των κρατών μελών. Ήδη με μεγάλες προσπάθειες εργοδός ε, προσπαθούν τα κράτη-μέλη να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Έχετε τρία λεπτά ως όριο στην παρέμβαση. Λυπούμε πολύ λέει ο μιλητή που ξεπέρασα τον χρόνο. Το τελευταίο αναφέρθηκε ότι είχαμε σε σχέση με την Ευρωζώνη αναφέρθηκε το ότι θα κατέρε λέει σε πέντε χρόνια. Βλέπουμε ότι σε σχέση με το πρότυπο το οποίο μπορεί να ακολουθηθεί δεν είναι οι καλύτερες προοπτικές αυτές. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπατε όπως και οι παρεμβάσεις των άλλων αγοριτών. Παρακαλώ όμως να τηρείτε το χρόνο. Σας ευχαριστώ ο συνάδελφος από την ε, ε, Ρουμανία, από την συνέλευση της ε, Ρουμανίας θα λάβει τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω... Ευχαριστώ. ήθελα να μιλήσω για τις ανανεώσιμες ενέργειες και να τονίσω ένα θέμα το οποίο ανέφερε ε, η κυρία Χάντσερ όσον αφορά την διαφοροποίηση πηγών ενεργείας και την καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών. Από πολιτικής απόψεως χρειαζόμαστε μία συμφωνία στον ενεργειακό τομέα που να αποτελέσει τη βάση για την εξάλληψη των μονοπωλίων και να αποφύγει τις ε, κρίσεις ε, που ζήσαμε στον τομέα του φυσικού αερίου. Χρειαζόμαστε όσο είναι γνωστόν απόθεμα. Το απόθεμα αυτό μπορεί να καταρτίζεται από κοινού από διάφορες χώρες. Η κυρία Χέντσερ ανέφερθηκε εις ε, την ε, ε, ηλιακή ενέργεια που μπορεί να αναπτυχθεί πολύ και στο Βόρειο Ευρώπη της αιωλικής ενεργείας. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει ένα, ένα πλαίσιο νομοθετικό για να προωθηθούν αυτές οι δράσεις και για να υπάρξει συγχρόνως μείωση κατανάλωσης ενέργειας Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Κλοντ Τούρμες, ε, Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι προκλήσεις είναι τεράστιες, διότι 85 έως 95% των μειώσεων που προβλέπονται μέχρι το 2050 απαιτούν μία αναδιάρθρωση όχι μόνο της ενεργειακής παραγωγής αλλά και των υπολείπων υποδομών. Άρα αυτά τα οποία αναφέρονται μέχρι στιγμής περιορίζονται στο πετρέλαιο και αρχίζουν ε, οι υπεύθυνοι της ασφαλείας στην Αμερική να ανησυχούν ήδη για την επάρκεια του πετρελαίου το 2015. Ε, άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, οποίες ενδέχεται εμείς να μην έχουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο έναυσμα για την ενεργειακή μας πολιτική. Έχω τρεις συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις ή του συντάξαντες στη μελέτη. Όταν μιλάμε για την πολιτική ε, αποβλήτων διότι μιλήσαμε ε, για την ε, ανακύκλωση και παραγωγή προϊόντων που δεν είναι επικίνδυνα. Δεν είδα όμως μία αρχίση, δηλαδή εάν η αποτελεσματικότητα και η ζήτηση βρίσκονται στην αρχή. Επίσης είχαμε διαπραγματευτεί σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρξει ένα ε, νέο ρυθμιστικός οργανισμός αλλά μας είχε περιορίσει περίπτωση Μερώνη. Ε, εάν λοιπόν ε, πρέπει να δούμε αν θα μπορούμε να ε, ξεπεράσουμε αυτά τα νομικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και επίσης θα ήθελα να ξέρω όσον αφορά τις συμφωνίες για την προμήθεια του αερίου εάν μπορούμε σαν Ευρωπαίοι να προχωρήσουμε διότι μειώνουμε την θέση μας έναντι π.χ. της Ρωσίας εάν κάθε μέρα έρχεται και χτυπά την πόρτα της Gazprom και του κυρίου Πούτιν ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό κράτη, κράτος. Ενώ εάν ήμασταν ενωμένοι ίσως θα είχαμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα λοιπόν να το σχολιάσετε αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ράινερ Βίτμαν της Αυστριακής Εθνικής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προμήθεια ενεργείας πρέπει ε, να ε, είναι εφικτή και να ε, εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Πρέπει να είμαστε πιο ασφαλείς για να ενισχύσουμε και την κοινή μας Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα διότι μιλάμε πολύ για την Ευρώπη των πολιτών αλλά όσον αφορά την προμήθεια ενεργείας αντιλαμβάνομαι ότι δεν προχωράμε χωρά κανείς επαρκώς. Ε, ατομική ενέργεια, 3% της ενεργείας ε, ε οφείλεται εις ε, την ατομική ενέργεια και ακούω πολλούς που τη συζητούν. Βέβαια ξέρω ότι υπάρχουν θέματα που δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη στα διάφορα κράτη, αλλά θα μπορούσε κανείς να αντικαταστήσει την τις ορυκτές πηγές ενέργειας αλλά υπάρχουν και ε, πηγές σαν το ουράνιο που είναι επικίνδυνες και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Αλλά ε, εμείς που δεν είμαστε ατομική χώρα ή Αυστρία συμβάλλουμε με ένα δισεκατομμύριο το χρόνο στο Ινευρατόμ Δεν θα ήταν λοιπόν καλύτερα να αποσύρουμε αυτά τα χρήματα και να τα χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού για να προωθήσουμε την Ευρώπη για τις ανανεώσιμες ενέργειες γιατί εμείς που δεν είμαστε ατομική χώρα γιατί πρέπει να συμβάλλουμε στο Ευρατόμ. Ευχαριστώ κύριε Βίτμαν και τώρα ο τελευταίος ομιλητής είναι ο Αντώνιο Κορέα Κάμπος. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ε, ξεκινήσω συγχαίροντας ε, τους ε, εθνικούς βουλευτές, τους συναδέλφους και τους αγορητές που ξεπώνησαν μια εξαιρετική έκθεση το να δημιουργήσουμε μια ενεργειακή κοινότητα που είναι επί της ουσίας η πρόταση της έκθεσης εξαρτάται από τις σημερινές επίκαιρες καταστάσεις, το πλαίσιο που δημιουργείται σε κάθε κράτος μέλος. Οι καταστάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από γεωγραφικές διαφορές που είναι σημαντικές. Έχουμε εξωτερικές εξαρτήσεις που είναι διαφορετικές. Έχουμε συνήθειες ενεργειακής κατανάλωσης που και αυτές είναι διαφορετικές. Πολιτικές τιμών πάλι διαφορετικές. Και η φύση των αγορών που ε, και αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και φυσικά εθνικές στρατηγικές. Υπάρχουν ε, στρατηγικές ε, που έχουν ε, ε, στρατηγική ανεξαρτησία, άλλες που έχουν στρατηγική συνεργασία. Εδώ η σύγκριση με την ΑΕΚΑΧ, με την κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα στην ΕΚΑΧΑ, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, υπήρχε γεωγραφική εγκύτητα των χωρών μελών παραγωγών. Υπήρχε τεχνολογικά μόνο μία μέθοδος παραγωγής και υπήρχαν αναδυόμενες ε, ε, δυνάμεις ε, όσον αφορά την αγορά που πίεσαν για να δημιουργηθεί αυτή η κοινότητα. Η κατάσταση είναι διαφορετική από εκείνη σήμερα. Παρόλες τις στρατηγικές και τις προτάσεις που παρουσιάζονται, είναι μια δυνατότητα ενδιαφέρουσα όλους τους λόγους. Πρώτα απ' όλα είναι ελαστική. Επιτρέπει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα να δραστηριοποιηθεί. Επίσης έχει τη δυνατότητα για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων. Όμως ενέχει κινδύνους. Έχουμε ε, και ε, τις ε, γεωγραφικές θα έλεγα συνιστώσεις και τα διαφορετικά συμφέροντα, τα διαφορετικά επίπεδα όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα των διαφορετικών χωρών και τις περιφερειακές στρατηγικές. Το ερώτημα που θέλω να διατυπώσω και ολοκληρώνω είναι πώς θα δημιουργήσουμε την κριτική, κρίσιμη μάζα αυτή για μια ενεργειακή κοινότητα του μέλλοντος που σιγά σιγά θα μετατρέπει μια εθελοντική, εθελούσια κοινότητα σε μια κοινότητα στραμμένη προς το μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Βουλευτά. Και τώρα στη συνέχεια Θα ακούσουμε τους ε, ειδικού μας, την κυρία Χάντζερ και τον κύριο Φαντεβότερ, να απαντήσουν στις, ε, που θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν θα είναι εύκολο να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Ίσως κάποιες γενικές παρατηρήσεις και στη συνέχεια η συνάδελφος Χάντσερ να απαντήσει σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα όπως αυτά που έθεσε ο κύριος Τούρμες. Καταρχήν, όσον αφορά την συνθήκη ΕΚΑΧ. Δεν είπαμε στην έκθεσή μας ότι η σημερινή η καλύτερη κατάσταση, μάλλον ότι η κατάσταση σημερινή οφείλεται στην ΕΚΑΧΑ. Είπαμε ότι τα νομικά μέσα που, κράτη, που είχαν τα κράτη-μέλη στη διάθεσή τους υπό τη συνθήκη ΕΚΑΧ ήταν ευρύτερα από αυτά που έχουν τώρα στη διάθεσή τους. Δεύτερον, υπάρχει ένα αίσθημα το οποίο δεχτήκαμε, είναι ένα αίσθημα κρίσης. Ε, εξαρτώμαστε από ε, τρίτα ε, κράτη για την ενέργεια. Αλλά υπάρχει και ένα θετικό στοιχείο σε αυτό το σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε. Αν αυτή η διαδικασία προς μια νέα κοινότητα ή μια πραγματική ενεργική πολιτική γίνει, θα υπάρχουν ευκαιρίες που θα καταστήσουν την Ευρώπη ε, χώρο εχμής για θέματα ενέργειας και άρα και βιομηχανικής εξέλιξης. Αυτά ως εισαγωγικές παρατηρήσεις. Επίσης θα ήθελα να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις. Καταρχήν, ακούσαμε μια αντίσταση σε σχέση με μια νέα συνθήκη. Όντως έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας και αν κατάλαβα καλά η συνθήκη της Λισαβόνας ακριβώς υπάρχει διότι περιλαμβάνει διατάξεις και ε, για θέματα ενέργειας και για, θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε αυτά και για να τα εκμεταλλευτούμε χρειάζεται πολιτική βούληση, το είπατε. Βούληση πολιτική όμως που σπανίζει και οι αντιλήψεις είναι διαφορετικές από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Γι' αυτό και προτείνουμε αυτή τη μικρή συνθήκη που βασίζεται στο πρότυπο Σέγγεν και που θα επιτρέπει σε ομάδες χωρών να προχωρήσουν ας πούμε όπως με την Βαλτική Πρωτοβουλία όπου οι χώρες της Βαλτικής προχωρούν σε μια μικρή ομάδα θα μπορούσαν να το κάνουν και οι σκανδιναβικές χώρες η Πολωνία, οι χώρες Βίσεγκρατ και εκεί γίνονται πρωτοβουλίες θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο μοντέλο για να μπορέσουν όλοι μαζί να προχωρήσουν σε, στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης ολοκλήρωσης και με σεβασμό στο κοινοτικό κεκτημένο υπήρχε και το θέμα των χαμένων και των κερδισμένων Πιστεύω πως εάν πρότυπο είναι τελείως εθελοντικό, ανάμεσα δηλαδή στα κράτη που το επιθυμούν, δεν υπάρχει κίνδυνος να μείνουν μερικοί χαμένοι και μερικοί να βγουν κερδισμένοι. Βασίζεται η συνεργασία στην βούληση των κρατών μελών να συμμετέχουν σε αυτήν. Τρίτη παρατήρηση για την ε, ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης χωρίς να θέλω να ε, παραστήσω τον ε, τεχνικό ή τον ειδικό, είμαστε νομικοί ειδικοί Μπορούμε ότι ε, μια εξέλιξη μπορεί να υπάρχει αν υπάρχει μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική που θα είναι προσανατολισμένη προς την έρευνα, προς μια κοινωνία χωρίς ε, διοξείδιο του άνθρακα θα μπορούσαμε να είμαστε να είμαστε αυτάρκεις όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προς τα αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Τέταρτη παρατήρηση και τελευταία. Σε όλα όσα άκουσα, πιστεύω πως σε μια ενεργειακή κοινότητα που θα βασίζεται σε ένα κοινό δίκτυο, είναι ασφαλής ε, ε, προσπάθεια, δηλαδή δεν θα έχουμε ε, αντίθετα αποτελέσματα αν συνδέσουμε όλα μας τα δίκτυα και τα συνδυάσουμε και αν δημιουργήσουμε έτσι μια πραγματική αλληλεγγύη. Δηλαδή, με βάση το Σέγγεν, το πρότυπο Σέγγεν και προς την κατεύθυνση της Κομισιόν θα ήταν μια επιλογή όπου δεν, υπάρχει.